πλησιάζουν οι γιορτές, ελπίζω οι διακοπές αυτές και η συμβολική αυτή περίοδος θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε στη δουλειά μας για τις απαλλαγές και πρέπει να βιαστούμε λίγο γιατί λόγω των εκλογών έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας από ό,τι κανονικά. Δεν έχουμε το χρόνο ιδιαίτερα για θέματα όπως συναντήσεις με επιτρόπους λοιπά. Λοιπόν, θέλετε να αλλάξει κάπου η ημερήσια διάταξη. Όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι η συνεδρίασή μας είναι μια δημόσια συνεδρίαση. Αναμεταδίδεται δικτυακά. Θέλω εδώ να καλωσορίσω και τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως επίσης και ε, τον Επίτροπο Τσίολος. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Είναι τα πρακτικά της συνεδριάσεως του μηνός Νοεμβρίου. Δεν υπάρχει κάτι εδώ. Και περνάμε στην απαλλαγή 2012 με εισηγητή τον κύριο Πίπερ. Έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Τσίολος. Επαναλαμβάνω. και θα του δώσω το λόγο αφού ακούσουμε τα εισαγωγικά σχόλια από πλευράς του Μάρκους Πίπερ, εφόσον θέλει το λόγο βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε κρατήσει ένα σχετικά καλό ρυθμό. Χρονικά έχουμε προχωρήσει αρκετά και θα ήθελα να κάνω λίγα σχόλια έτσι ώστε να δώσω τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει σε, στα ίδια θέματα. Κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ξέρετε ότι η γεωργική οικονομία είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα πιο μεγαλύτερα κομμάτια του κοινοτικού προϋπολογισμού και είναι και κάτι το οποίο προκαλεί γενικότερα την προσοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Ενδιαφέρονται οι Ευρωπαίοι πολίτες για την γεωργική οικονομία. Ε, θα μιλήσουμε για τον πρώτο πυλώνα καταρχάς και δεύτερον θα παρουσιάσω τα υπόλοιπα θέματα. Κάτω από τον πρώτο πυλώνα λοιπόν έχουμε ένα ποσοστό λάθος 2,9% μετά από το 3,8% ε, που είχαμε σημειώσει πέρυσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ε, ε, είναι κάτι που το συζητάμε για πρώτη φορά και υπάρχουν πολλές αιτίες για, αυτού το, για αυτό το ποσοστό λάθους. Έχουμε τώρα ένα νέο σύστημα εντοπισμού το LPIF, στο οποίο θα αναφέρομαι ε, αρκετά μετά, και το σύστημα αυτό λειτουργήσε εν μέρη φέτος. Το συνέδριο επισκέφθηκε κάποιες, ε, ε, εξέτασε το θέμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λουξεμβούργο και εμείς ασχοληθήκαμε με άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και Να πω ε, για την Πορτογαλία ότι οι επιφυλάξεις για το LPIF βασίστηκαν στα πρώτα στοιχεία που είχαμε συλλέξει το 2007. Και δεν μπορούμε να πούμε το 2013 πως ε, έχουν ε, αρθεί τελείως οι ε, επιφυλάξει μας αυτές ε, θα δούμε θα γίνει το 2015-2016 10 χρόνια δηλαδή μετά την πρώτη διαπίστωση των ε, λήψεων στη Γαλλία επισημάνθηκαν οι πρώτες ελλείψεις το 2007 και η Κομισιόν το 2013 είπε πως η Γαλλία θα έπρεπε να διορθώσει τον έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις μη συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Καταρτίστηκε το 2013 ένα σχέδιο δράση και εκεί πέρα θα έχουμε αποτελέσματα το 2013, 2015 ε, με για λήψεις που επισημάθηκαν πρώτη φορά το 2007 στην ε, Βουλγαρία. Βεβαίως η Βουλγαρία ε, είναι νέο κράτος μέλος αλλά το σύστημα εκεί πέρα έχει πρόβλημα και για αεροφωτογραφίες. Μια υπόθεση η οποία 2014-2015 θα ε, έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά τα πράγματα έτσι απλά. Η Κομισιόν τουλάχιστον στην ε, γεωργική πολιτική έχει τη δυνατότητα μέσω των αιτήσεων εκθέσεων να επιβάλλει αιτήσει διορθώσεις. Αλλά και εδώ πέρα ανησυχούν πάρα πολύ για την διάρκεια αυτής τη διαδικασία. Στη Γαλλία η διαδικασία αυτή ε, ολοκληρώθηκε το 2013 για το 2008. Με την Πορτογαλία θα κλείσουν οι λογαριασμοί του 2009-2011 μέχρι το 2014 και αυτό κρατάει χρόνια και συνολικά η διαδικασία δεν είναι και πολύ διαφανής δυστυχώς. Για εμάς ως εξωτερικούς είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε μήπως είναι απλούστερο να κάνουμε μια διόρθωση κατά για όλα τα στήματα που δεν λειτουργούν ε, πλήρως και χωρίς προβλήματα κρίνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο μου συγχωρείτε. Ε, κάθε φορά έρευνα διαφορετικές χώρες αλλά σε όλες βρίσκει σοβαρές ε, λήψεις και όσον αφορά αυτό το σύστημα το, το LPTS αλλά πάντα λέγανε πως ε, θα αλλάξουν τα πράγματα, θα διορθωθούν, αλλά πλέον ε, έχουμε την αίσθηση πως ε, η Κομισιόν υποτιμά την σοβαρότητα της κατάστασης. Να είπαν και για το όριο σημαντικότητας. Ελπίζουμε πως θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αλλά τι σύσταση μπορείτε να δώσετε εσείς ε, σε έναν εισηγητή ο οποίος ε, πρέπει να δώσει απαλλαγή, να πει ένα ναι ή όχι. Δύσκολα τα πράγματα. Και εδώ πέρα με τους συναδέλφους συμφωνούμε πως οπωσδήποτε πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα για ένα αποφασισμό. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα, ε, και εκεί το ποστό σφάλματος από το 7,7 ανέβηκε στο 7,9% ε, εδώ πέρα μιλάμε για τον ΦΠΑ, για τις δημόσιες προμήθειες και το συνέδριο στον δεύτερο πυλώνα διαπίστωσε προβλήματα σε Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Πριν από αυτό ήταν η Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Φιλανδία. Πριν από αυτό πάλι κάποιες άλλες χώρες μέχρι να αποκτήσουμε όλο το σετ. Έτσι οπότε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από ό,τι φαίνεται στην εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα αν εμπιστευτούμε το ελεγκτικό συνέδριο που το εμπιστευόμαστε. Η ΔΕ Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, είχε μια γενική επιφύλαξη στην ετήσια έκθεση για 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στο δεύτερο πυλώνα. Ε, μεγάλα ποσά. Εδώ πέρα λοιπόν αναμένουμε κατεπηγόντως βελτιώσεις και έρχομαι τώρα στο τέλος να συνοψίσω. Συνολικά έχουμε την εντύπωση πως το σύστημα δυστυχώς δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται. Ο δεύτερος πυλώνας έχει τον δεύτερο το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων από όλες τις πολιτικές και στον πρώτο πυλώνα ε, εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλα προβλήματα για την καταγραφή των εκτάσεων, κατά το οποίο δεν έχει λυθεί και μας λένε πως τα πράγματα που ξεκίνησαν τώρα θα αποδώσουν 2015-2016. Ε, Αυτά λοιπόν για τις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Χτες ακούσαμε πως ε, στον τομέα των καθαρών διορθώσεων πρέπει να ε, καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά νομίζω πως ειδικά στον τομέα της γεωργίας πραγματικά έχουμε τεράστιες προκλήσεις. Και αναμένω τώρα να Ακούσα τη συζήτηση με επίτροπο και ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Είναι καλό το ότι έχουμε εδώ πέρα τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι τόσο σημαντικό ο προπολογισμό της Γεωργίας ώστε έχουμε σήμερα δύο μέλη του ελεκτικού συνεδρίου, η κυρία, ο κύριος Κουμπίκ και η κυρία Κούτπερτ. Ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Κουμπίκ. Dear Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της προσπάθειας που έχει κάνει το ελεγκτικό συνεδρίο στα πλαίσια της αξιολόγησης της άμεσης στήριξης και της λειτουργίας της γεωργική αγοράς. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τον πρώτο πυλώνα. Στις πληρωμές 3,8% είναι το ποσοστό λάθους. Εμείς χρησιμοποιούσαμε 180 δείγματα και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα εν μέρη ε, βρέθηκαν αποτελεσματικά. Αυτά είναι τα γενικά συμπεράσματα μετά από την εξέταση ε, πέντε ευρύτερων περιπτώσεων. Θα σας δώσω ίσως κάποια, περι, κάποια περισσότερα στοιχεία. Τι είδους λάθη έχουν συνεισφέρει σε αυτού του είδους ε, το ποσοστό, σε αυτού του ύψους το ποσοστό λάθους. Καταρχάς για τις δηλώσεις γης ε, υπήρξαν προβλήματα. Έχουν κάποιοι δηλώσει περισσότερη ε, γη και επίσης έχουν δηλωθεί και πληρωθεί και περιοχές οι οποίες δεν ήσαν επιλέξιμες. Άλλα λάθη αφορούν κάποιες λανθασμένες αποφάσεις από πλευρά των κρατών μελών. Τα προβλήματα αυτά είναι υπεύθυνα για πάνω από το 1 τρίτο του MLE. Τα υπόλοιπα λάθη προέρχονται από διάφορες, ε, διάφορα προβλήματα όπως επίσης ε, και θέματα πολλαπλής συμμόρφωσης επίσης. Αν συγκρίνουμε τώρα το 2011 με το 2012 και τα ποσοστά λάθος, βλέπουμε ότι οι αριθμοί εξηγούν από μόνοι τους το πως έχει η κατάσταση. Το ποσοστό λάθος ανέβηκε από το 2,9 στο 3,8 με το ανώτατο όριο στο 5,9 και το κατώτερο στο 1,7. Όμως βλέπουμε αρκετές αναλογίες εδώ με το 2011. Η συχνότητα αυξήθηκε ε, πολύ λίγο, το πως, ο αριθμός των ε, ποσοστοποιήσιμων λαθών αν θέλετε παραμένει ο ίδιος Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και ποσοστά λαθών, ε, κυρίως διοικητικά λάθη ε, και η πολλαπλή συμμόρφωση, τα λάθη στην πολλαπλή συμμόρφωση είναι το 0,2%. Είναι θέματα που αναλύσαμε, τα δεδομένα τα αναλύσαμε και είδαμε ότι έχουμε περισσότερα μεγάλα λάθη το οποίο μαθηματικά εξηγεί την αύξηση του ποσοστού. Νομίζω ότι ο λόγος, επιμέρους τουλάχιστον λόγος αφορά, που δημιουργήθηκε η κατάσταση αυτή είναι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων, κάτι το οποίο με οδηγεί στο επόμενο τμήμα της αξιολόγησής μου. Τώρα, σε επίπεδο κρατών μελών, η αξιολόγηση του συστήματος. Εμείς, σαν ελεγκτικό συνέδριο, σε αιτήσια βάση ελέγχουμε ορισμένες χώρες και καταλήξαμε σε κάποια αρνητικά συμπεράσματα. Ε, η αποτελεσματικότητα του IACS επηρεάζεται από ανακριβή στοιχεία. Δεύτερον, το συνέδριο έχει επαναλάβει έναν αριθμό επιμέρους μετρήσεων από, τους, από τις υπηρεσίες πληρωμών μετά από τις επιτόπιες ε, έρευνες και σε τρία κράτη-μέλη οι μετρήσεις μας οι μετρήσεις μας ήταν διαφορετικές από αυτά από αυτές τις οποίες μας είχαν δηλώσει. Βρήκαμε επίσης ότι το σύστημα που λειτουργεί για τη διαχείριση της βοήθειας ε, ε, στα πιο ευάλωτα πρόσωπα στα διάφορα κράτη-μέλη να ε, λειτουργήσε αποτελεσματικά. Αλλά για έναν μεγάλο αριθμό συναλλαγών που επηρεάζονται από λάθη, το συνέδριο θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές είχαν αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να ανοιχνεύσουν σωστά και να διορθώσουν τα συγκεκριμένα λάθη. Αυτά ήταν τα λάθη σε επίπεδο κράτης μέλους, σε επίπεδο τώρα επιτροπής. Στην ετήσια έκθεσή της ε, για το 2012 η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έκανε μια αναθεώρηση στον υπολογισμό του ποσοστού λάθους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές των επιθεωρήσεων που έγιναν στα κράτη-μέλη και που εστάλησαν από τα κράτη-μέλη επηρεάζονται από την αναξιοπιστία τους ή μάλλον από την έλλειψη αξιοπιστία τους. Έτσι λοιπόν το ποσοστό λάθους για τις αποσυνδεδεμένες περιοχές για το 2012 υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι 2,4%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι στο, στη μέση του χαμηλότερου και του υψηλότερου ορίου όπως υπολογίστηκε από το συνέδριο ε, για το σύνολο 1,7 με 5,9. Παρουσιάζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά θα περάσω τώρα στις συστάσεις. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των στοιχείων εμείς ε, προτείνουμε ότι η επιλεξιμότητα των γεών είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται σωστά στο LPIS. Πρέπει να υπάρξει άμεση δράση σε επίπεδο διοικητικό και ελεγκτικό και σε επίπεδο... Payments Σε επίπεδο Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρξουν πληρωμές που να βασίζονται στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Και τέλος η σχεδίαση και η ποιότητα των εργασιών ε, των διευθυντών των υπηρεσιών πληρωμών και των σωμάτων πιστοποίησης θα πρέπει να παρέχουν μια αξιόπιστη βάση που να διασφαλίσει το τακτό ε, των ε, παρεμβάσεων αυτών. Τώρα, κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η τροποποίηση της τάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τον υπολογισμό του ποσοστού λάθους είναι ένα καλό βήμα. Η νέα αντιμετώπιση δεν είναι κάτι το οποίο έχει υποστεί ε, λεπτομερή έλεγχο αλλά θεωρώ ότι είναι καλό που έχει λυθεί το συγκεκριμένο βήμα και ελπίζω να συνεχιστεί η βελτίωση. Δεύτερον θα ήθελα να υπογραμμίσω την σωστή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες του Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως φαίνεται και από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από αυτά που είδαμε στα πλαίσια των συναντήσεων που κάναμε είναι ότι δεν διαφέρουμε ε, πάρα πολύ σε σχέση με την αξιολόγηση της φύσης των προβλημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Κούμπικ που μας παρουσιάσατε την εκθέση από την πλευρά του συνεδρίου και δίνω το λόγο στην κυρία Κούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 4 της της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου που, αναφορά, που αναφέρεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, την αλληλεία και την ε, υγεία. Αυτές οι περιοχές καλύπτουν το 10% του ευρωπαϊκού προπολογισμού για το 2012, δηλαδή 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέντε κυρία σημεία θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο της εκθεσής μας. Πρώτον, υπήρχε σημαντικό πραγματικό ύψος φάλματος. Το πλέον πιθανό σφάλμα ανήλθε στο 7,9% δηλαδή πολύ κοντά στο περσινό, στην περσινή τιμή. Το 195% το περιθώριο ε, ε, εμπιστοσύνης βρίσκεται μεταξύ 4,5% και 11,3% για το ποσοστό σφάλματος. Επίσης διαπιστώσαμε προβλήματα στα 2 τρίτα των πληρωμών στους οποίες ασκήσαμε έλεγχο, το οποίο σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ε, πολύ διαδεδομένο. Διαπιστώθηκαν προβλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη και μάλιστα σε όλα τα μέτρα ενίσχυσης τα οποία ε, υποβάλαμε σε έλεγχο. Δεύτερο σημείο. Κατά την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να έχουν ε, εντοπίσει και να έχουν διορθώσει την πλειονότητα αυτών των σφαλμάτων. Τρίτον, οι δικαιούχοι δεν ε, σεβάστηκαν τις ε, απαιτήσεις επιλεξιμότητας, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας παραμένουν περίπλοκες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Αλλά επίσης και εξαιτίας ελλείψεων στα συστήματα των κρατών μελών. Τα κύρια προβλήματα εμφανίστηκαν όταν δεν εφαρμοστήκαν σωστά οι κανόνες περί δημοσίων συσβάσεων, όταν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα δεν εφαρμόστηκαν ή δεν έγιναν σεβαστά και οπουδήποτε επελέγησαν και χρηματοδοτήθηκαν έργα ή δικαιούχοι οι οποίοι δεν ήταν επιλέξιμοι. Επίσης, το 1 τρίτο των περιπτώσεων των σφαλμάτων ε, οι υποθέσεις συνδέονταν με ε, προβλήματα πολλαπλής ε, συμμόρφωσης. Τέταρτον, το συνέδριο αξιολογεί τα συστήματα ελέγχου ως μερικώς αποτελεσματικά, όχι πλήρως αποτελεσματικά. Πέμπτον, το συνέδριο συνιστά στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν όλες τις ε, πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Κάτι που θα τους επιτρέψει να εντοπίσουν και να διορθώνουν την πλειονότητα των σφαλμάτων. Και θέλω να είμαι σαφής δεν ζητάμε περισσότερους ελέγχους, ζητούμε οι έλεγχοι που ήδη προβλέπονται να εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά από το κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελληνικού Ελεκτικού Συνεδρίου για την απαλλαγή του 2012 που καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή των ε, υφιστάμενων κανόνων παραμένει μη ικανοποιητική. Επίσης όσον αφορά την αποδοτικότητα και εδώ η κατάσταση δεν είναι ε, καλή. Γιατί τίθενται στόχοι οι οποίοι είναι προβολικά γενικο, γενικοί. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα έργα δεν καταλήγει τελικά στην επιλογή των βέλτιστων έργων και δεν υπάρχει ε, μια σαφής κατεύθυνση στην ε, χρήση αυτών των δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Περισσότερε πληροφορίε για τα ζητήματα αυτά μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 10 τη ετήσια μα έκθεση. Ε, Κοιτώντα ε, συγκριτικά τα συμπεράσματα του κεφαλαίου 4, θεωρούμε ότι χρειάζεται να συνεχιστεί ε, ο έλεγχος, ο επισταμένος έλεγχος του τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειάζονται νέα προγράμματα δράσης στη νέα προγραμματική περίοδο, τα νέα προγράμματα δράσης και η προσπάθεια απλοποίησης ίσως ε, επιλύσει κάποια από τα προβλήματα. Παρόλα αυτά παραμένει υψηλό επίπεδο κινδύνου σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στα ε, μέτρα ε, χρηματοδοτικής ε, μόχλευσης. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχουν με τρόπο προσεκτικό τον τομέα αυτό, η Επιτροπή, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και το Ελεκτικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τις εισαγωγικές παρατηρήσεις των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Καταρχάς θα αναφερθώ σε τρία μέτρα τα οποία συνδέονται με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Στις 12 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε νέες διορθώσεις 305 εκατομμυρίων. Αυτό οδηγού, οδηγεί σε 1,3 δις διορθώσεων οικονομικών. Όπως όλες αυτές οι διορθώσεις είναι καθαρές διορθώσεις τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από τα κράτη-μέλη για άλλους στόχους. Τα χρήματα αυτά χάνονται δηλαδή για τα κράτη-μέλη τα οποία έκαναν λάθη. Οι καθαρές αυτές διορθώσεις δεν είναι μόνο μία μορφή προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά και κίνητρο για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισής τους. Δεύτερον, οι πρόσφατες αλλαγές του κανονισμού σε σχέση με τη διακοπή πληρωμών λόγω της λειτουργίας των ελεγκτικών συστημάτων μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα διακοπής για ένα περιφερειακό πρόγραμμα στην Ιταλία, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Τον Ιανουάριο του 2014 τα νέα γενικά καθεστώτα διακοπής πληρωμών που προήλθαν από τη μεταρρύθμιση του ΚΑΠ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Αυτό που κάναμε φέτος λοιπόν είναι με την ισχύουσα νομοθεσία την οποία βελτιώσαμε πέρυσι και με τους νέους κανόνες νομίζω από το 2014 θα χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μέσα με πιο αποτελεσματικό τρόπο και αρκετά ενωρίς. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν μέρη ε, ε, κατάργησε το μνημόνιο σε σχέση με τις εξαιρέσεις για την Ελλάδα γιατί οι τοπικές οι εθνικές αρχές δεν είχαν θέσει σε λειτουργία ένα τμήμα των προγραμμάτων δράσης έτσι ώστε να συνεχιστεί η, ε, το μνημόνιο, η ισχύ του μνημονίου. Οπότε η Ελλάδα θα μπει στο κανονικό καθεστώς από τον Ιανουάριο του 2014. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα προστασίας του προϋπολογισμού της Ένωσης που λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο στην ΚΑΠ. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε όπως είπατε να έχουμε ένα, ένα ποσοστό λάθος μη ικανοποιητικό και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Για τον πρώτο πυλώνα το ποσοστό λάθους που εντοπίστηκε από το συνέδριο είναι υψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Διαπιστώνει όμως η ίδια, το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο το ένα μεγάλο τμήμα των σφαλμάτων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή διορθωθεί από πλευρά των ιδίων των κρατών μελών. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το, το ως, δε, ως σύστημα αλλά η ποιότητα της διαχείρισής του από τα διάφορα κράτη-μέλη. Εμείς προκαταλάβαμε αν θέλετε τα συμπεράσματα του συνεδρίου βελτιώνοντας τις μεθόδους υπολογισμού ε, των ε, σφαλμάτων και για τα μέτρα των αγορών. Ε, εντοπίσαμε τρία κράτη-μέλη, τα είπατε άλλωστε, η Πορτογαλία, Βουλγαρία και Γαλλία και είπαμε ότι αυτές οι τρεις χώρες έχουν οδηγήσει κυρίως στην αύξηση αυτού του ποσοστού λάθους. Για τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει ήδη προγράμματα δράσης και το πρόβλημα, τα προβλήματα που υπήρχαν με το LPIS βρίσκονται σε φάση επίλυσης. Το 2014 θα γίνει έλεγχο στη Βουλγαρία για την ε, αξιολόγηση της ποιότητας του LPIS Στη Γαλλία δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα δράσης πιο περίπλοκο και κάποιες οικονομικές διορθώσεις έχουν ήδη επιβληθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Πέρα από αυτά τα τρία κράτη-μέλη, ένα οριζόντιο πρόγραμμα δράσης που καλύπτει το καθεστώς των άμεσων πληρωμών θα τεθεί σε λειτουργία. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας για να εμβαθύνουμε καλύτερα στις βασικές αιτίες σφάλματος. Ε, στο μέλλον λοιπόν θα ενισχύσουμε την ικανότητα πρόληψης εκ των προτέρων και συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Δημιουργήσαμε στο εσωτερικό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας μια νέα μονάδα για την παρακολούθηση της εξέλιξης των άμεσων πληρωμών και θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου του 2014 για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το επίπεδο σφάλματος είναι περίπου το ίδιο με τον προηγούμενο χρόνο. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει ήδη πολλαπλές δράσεις και θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, όπως άλλωστε έχουμε αναφέρει ήδη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά όμως απαιτούν χρόνο και τα αποτελέσματα θα έρθουν αλλά σταδιακά λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου χαρακτήρα του πολιετού ε, που χρησιμοποιούμε στον προγραμματισμό μας. Πολλές χώρες μέλη απλοποίησαν τα προγράμματά τους σε σχέση με το τι είχαν κάνει πέρυσι και με το νέο προγραμματισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και θα απαιτήσει κάποια απλά και ελέγξιμα εύκολα κριτήρια επιλεξιμότητας. Να υπογραμμίσω ότι ένα ποσοστό λάθους 7,9% δεν σημαίνει ότι 7,9% του προϋπολογισμού χάθηκε. Όχι. Πρέπει ε, να πω ότι δεν υποτιμάμε το ποσοστό βέβαια αυτό του σφάλματος και ακόμα και αν ένα σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου δεν είναι συμβατό, μπορεί να προσφέρει ε, ε, επιπλέον αξία και να πετύχει το στόχο του. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην κοινή διαχείριση, μόνο μια κοινή δράση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είναι αποτελεσματική. Ε, το έχω πει στους Υπουργούς Γεωργίας επανειλημμένα και ελπίζω ότι τα μέσα μας ε, θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της διακοπής ε, και της πλήρους επίσης ε, διακοπής των πληρωμών, κάτι το οποίο θα δώσει περισσότερα μέσα στις εθνικές πολιτικές. Για τις οικονομικές διορθώσεις παίρνουμε επίσης μέτρα και ο κύριος Πίπερ πάρα πολύ σωστά υπογράμμισε τη μεγάλη διάρκεια της περίοδου αυτής. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι σύντομη. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις προθεσμίες που είναι 4 με 5 χρόνια σήμερα σε 2 χρόνια. Και με τις νέες οργανώσεις, τις νέες δυνατότητες οργανωτικές θα το πετύχουμε. Οι νέες ευθύνε ε, των οργανισμών πιστοποίησης επίσης στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, εθνικών μηχανισμών ε, πιστοποίησης θα ενισχύσουν ε, τους στόχους αυτούς αυτές οι υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τον νέο κανονισμό θα πρέπει να κάνουν ε, στατιστικά αξιόλογα δειγματολόγια τα οποία θα επιτρέπουν να εντοπίζουμε ακόμα και μεμονωμένες συναλλαγές. Εμείς σε επίπεδο τεχνικό και σε επίπεδο κατάρτισης θα συνοδεύσουμε την προσπάθεια αυτή έτσι ώστε οι μηχανισμοί πιστοποίησης να λειτουργήσουν σωστά. Από το 2014 στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ θα υπάρχουν διπλάσιες διαδικασίες ελεγκτικές και αποστολές σε σχέση με το 12. Και ο νέος πολιετής προγραμματικός χαρακτήρας ε, των ελέγχων ε, σε ένα σύστημα το οποίο στοχεύει στους συγκεκριμένους κινδύνους θα γίνει πιο αποτελεσματικό. Αυτό το μέσο λοιπόν το συντονισμένο και η συνεργασία με τους μηχανισμούς πιστοποίησης θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει επί τόπου και να βελτιώσουμε την ικανότητα παρέμβασή μας πριν από τις οικονομικές διορθώσεις. Ε, κατά τη διάρκεια της παρούσης εντολής είναι η τελευταία φορά την οποία παρουσιάζομαι εδώ την παρουσία του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι εμείς υπερασπιστήκαμε τα οικονομικά συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογούμενου και σε επίπεδο περιεχομένου και σε επίπεδο ωφέλους για την ΚΑΠ και σε σχέση με τις διορθώσεις, τον τρόπο χρήσης των χρημάτων που είχαμε στη διάθεσή μας. Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή ήταν καθοριστική. Πάρα πολλές από τις βελτιώσεις τις οποίες κάναμε, τις κάναμε χάρη στη δική σας στήριξη. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και υπολογίζω στη συνέχεια τη υποστήριξή σα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα ακούσαμε και το Ελληνικό Συνέδριο και τον Επίτροπο. Ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Πίπερ ζήτησε πάλι το λόγο. Όχι, όχι. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση. Κοιτάξτε, θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως του χρόνου θα κάνουμε τον απολογισμό. Μαθαίνω ότι θα κατέβεται και υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε αλλάζουν τα πράγματα, δεν θα είστε εκεί πάνω. Λοιπόν, Κοιτάξτε, ε, αυτό το οποίο μας δημιουργεί επιφυλάξει δεν είναι το ότι θεωρούν πως δεν αντιδρούν τα, τα μέσα προβλήματα, αλλά το πώς αντιδρούν. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα φέτος μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου του 2003 και τα προβλήματα είναι τα ίδια. Έτσι κοιτάξτε, δεν έχουμε φετίχ με το ποσοστό σφάλματος, αλλά είναι η κορφή του παγόβουνου και δείχνει το πώς λειτουργεί μια διοίκηση. Και μετά από αυτά τα οποία ε, μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο πριν από 10 χρόνια, φαίνεται πως δεν λειτουργεί καθόλου. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν με τη μη λειτουργία αυτή αφενός, ε, πάντα επί της αρχής έχει ελπίδα και λέει του χρόνου καλύτερα. Είτε με το νέο πολιτισμό πλαίσιο, με τη νέα διοίκηση, με το νέο οτιδήποτε. Εγώ πλέον έχω χάσει κάθε ελπίδα. Ε, δηλαδή η ελπίδα δεν βελτιώνει ε, τα πράγματα αυτά. Εντάξει, καθολική είμαι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να, να αρχίσουμε και εμείς να κουνάμε τα χέρια μας. Να μην ελπίζουμε μόνο. Κοιτάξτε, βλέπουμε εδώ πέρα επίση διαφορετική αντιμετώπιση των ιδίων πραγμάτων. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη για τα οποία γίνονται σχέδια δράση, για άλλα πάλι όχι. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι πώς υπολογίζετε το, το πόσο στο σφάλματος. Μία έχετε ένα επιπρόσθετο 2% αλλού έχετε ένα επιπρόσθετο 5%. Οπότε το ερώτημα είναι γιατί παραδείγματο χάρη για τη Βουλγαρία και την ε, Ρουμανία ε, επιφυλάξεις δικαίως για να αλλάξει κάτι και για τις χώρες παραδείγματος χάρη για τις οποίες, ε, τις οποίες αναφέρει το Ελληνικό συνέδριο από το 2007 Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, ε, Αυστρία γιατί δεν γίνεται τίποτα εκεί έχει σχέση με αυτό το οποίο λέτε το, το top-up. Γιατί σε άλλους υπάρχει αύξηση 2%, σε άλλους 5% και στο 5% ε, υπάρχει αντίδραση και στο 2% όχι. Συνεχίζετε κατάσταση και δεν κάνετε τίποτα. Προσπάθησα να το καταλάβω δηλαδή πραγματικά γιατί στον έναν γίνεται κάτι και στον άλλον όχι το θέμα του reputational risk με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εντάξει. Αλλά αυτό υπάρχει και για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία για πρώτη φορά αναφέρθηκε το 2007 από το ελεγκτικό συνέδριο. Το 2003 η έκθεση αναφέρει ήδη τα προβλήματα στην Ισπανία με το ότι δεν έχει υπάρξει διαχωρισμός του LPS ε, και τους βοσκοτόπους. Ε, επίσης αναφέρεται Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία χώρες οι οποίες έχουν μέχρι και σήμερα προβλήματα. Οπότε από πού προκύπτει αυτή η φοβερή υπομονή της Κομισιόν και η ελπίδα. Επίσης είπαμε σε άλλους ε, αύξηση 2% σε άλλους 5% και βέβαια κάποιοι ξεπερνάνε πιο εύκολα το, το όριο, το κατόφλι. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι όπως σας είπα γιατί αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα ίδια ή παρόμοια πράγματα. Μετά. Αυτό το οποίο είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν χρειάζονται περισσότερη έλεγχη αλλά καλύτερη έλεγχη. Αυτό είναι και το δικό μας το πρόβλημα εδώ και χρόνια και έχουμε όπως είπαμε 28 υπηρεσίες που κάνουν την καταμέτρηση και το, η ερώτηση 45 δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, τι έγινε με τους φορείς πιστοποίησης, ποια αποτελέσματα είχαμε. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω στο ερώτημα 34 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα και ποια μέτρα δεν επιτράπηκαν. Εγώ θα το παρακολουθήσω αυτό το ζήτημα, γιατί πάρα πολλές από τις ερωτήσεις οποίες θέσαμε απαντήθηκαν τελείως πρόχειρα. Ε, δεν έχουν απαντηθεί στην ουσία, έτσι, με την ακρίβεια που θα θέλαμε. Δηλαδή, όταν ρητάμε για προβλήματα, μας απαντάτε ποιο είναι το σύστημα. Μα το ξέρουμε ποιο είναι το σύστημα, για το πρόβλημα δεν μας λέτε τίποτα. Μετά, η διαδικασία διόρθωσης. Μα όταν ξεπερνάει τις χίλιες μέρες, ε, χάνεται οποιαδήποτε αξιοπιστία και, και νόημα στην ε, διαδικασία αυτή, έτσι. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν για να συντομεύσει αυτή η διαδικασία και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Μάλιστα σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Πολλές ερωτήσεις αλλά προτείνω να τις μαζέψουμε όλες μαζί. Μετά, ο κύριος Βόβεν. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συζητητές ήταν εξαιρετική η παρεμβασή του, καθώς επίσης και η παρέμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που μας θύμισε με την παρουσία του. Γνωρίζω ότι το ζήτημα των σφαλμάτων σας απασχολεί και προσπαθείτε να υιοθετήσετε μέτρα για να μειωθεί αυτό το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος και να ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα ήταν και η δημιουργία της μονάδας ε, ορκωτών ελέγχων. Άρα πράγματι το θεωρείται σημαντικό και το, το, το, το θέμα. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες ερωτήσεις, μια πιο γενική. Ξεκινώ από αυτή. Πρώτα απ' όλα τις καθαρές διορθώσεις. Γνωρίζουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Θεωρείτε ότι οι καθαρές διορθώσεις τελικά οδηγούν σε μείωση του σφάλματος. Θα ήταν χρήσιμο να το γνωρίζουμε αυτό όταν συζητάμε για καθαρές διορθώσεις και σε άλλα τμήματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Επίση θα ήθελα να γνωρίζω λίγα στοιχεία περισσότερα για τη μεθοδολογία που ακολουθεί το ηλεκτρικό συνεδρίο. Ο επίτροπο είπε ότι η μεθοδολογία του συνεδρίου, η αλλαγή τη μεθοδολογία, οδήγησε σε μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματο το 2012. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Γιατί. Επίσης, δύο ερωτήματα σχετικά με κράτη-μέλη. Πολλοί έχουμε εστιάσει στην ευθύνη των κρατών μελών για το πόσο για σφάλματος. Στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης ε, αναφέρομαι στην ε, ερώτηση 32, στην οποία ε, απαντάτε λέγοντας ότι πολλά κράτη-μέλη αναλαμβάνουν ε, συγκεκριμένες δράσεις ε, για την βελτίωση του συστήματος. Θα ήθελα ορισμένα παραδείγματα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα ε, βελτίωσης τη κατάσταση και επίλυσης των προβλημάτων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχία. Συγγνώμη, το το ΩΣΔΕ, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείριση και Ελέγχου. Όλοι θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο, το είπε και το Ελεκτικό Συμβούλιο, όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αλλά θα ήθελα να μα δώσετε ορισμένα παραδείγματα ε, κρατών μελών που αξιοποίησαν με σωστό τρόπο το ΆΙΕΚ, το ΩΣΔΕ. Ίσως η τεχνογνωσία των κρατών μελών που αξιοποιούν το ΩΣΔΕ να μπορούσε να μεταβιβαστεί και στα κράτη-μέλη που δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Ευχαριστούμε. κύριος Ευχαριστώ και σας καλωσορίζω, Επίτροπε Τσιόλος. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Είμαι λιγάκι μπερδεμένος όμως και παραμένουν, παραμένουν ορισμένα ερωτήματα. Δηλαδή, ως βουλευτής αναρωτιέμαι αν μπορώ να δώσω απαλλαγή. Γιατί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί Τη, με συγχωρείτε το, Ευρωπαϊκό, το Συνέδριο χρησιμοποιεί την έννοια του περιθωρίου του ποσοστού σφάλματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας παραπέμπω στην παραγραφό 10, απαντά διαφορετικά. Δηλαδή αναφέρεται στην ερώτηση 10 ότι το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκαν οι κανόνες δημοσίων συμβάσεων δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ε, αυξάνει το, ποσοστό ασφάλματος. Πώ είναι δυνατόν αυτό. Άλλο, ρωτάει, άλλο λέει το ελεκτικό συνέδριο, άλλο απαντά η Κομισιόν. Η Κομισιόν μας απαντά για περιπτώσεις απάτης και υπεξαίρεση χρημάτων, ενώ το ελεκτικό συνέδριο θέτει το ζήτημα του, ε, περιθωρίου, του ποσοστού σφάλματος. Δηλαδή το ερώτημα ήταν ότι το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος έχει ξεπεράσει ένα όριο και εσεί μα απαντάτε για το τι θα γινόταν σε περίπτωση επιξέρωσης χρημάτων. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τους ορκωτούς ελέγχους, έτσι ώστε να γνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Ε, ίσως να πρέπει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση, γιατί καταρχήν το δείγμα είναι εξαιρετικά μικρό. 180 ε, υποθέσεις και αναρωτιέμαι ποιο είναι το, το σύνολο των χρηματοδοτήσεων συνολικά. Όταν έχουμε χιλιάδες τέτοιες χρηματοδοτήσεις, να λαμβάνουμε ένα δείγμα 180 υποθέσεων μόνο, είναι εξαιρετικά μικρό, είναι εξαιρετικά προβληματικό κατά την άποψή μου. Δίνεται ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% στο δεύτερο τομέα των, της περιφερειακής ε, ανάπτυξης, αλλά είναι τεράστιο ε, το ποσοστό σφάλματος σε σχέση με αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν λέμε ότι το ποσοστό σφάλματος είναι 11% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% είναι τεράστιο το ποσό αυτό και το θέμα αυτό θα έπρεπε να αποσχολήσει σοβαρά την Επιτροπή. Πρέπει να ξαναδούμε τη μεθοδολογία τη στατιστική μεθοδολογία. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε το, ευρωπαϊκό το ελεγκτικό συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παράσχουν συγκεκριμένες εκθέσεις για συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα η πολλαπλή συμμόρφωση ή η ε, κοινή διαχείριση. Κύριε Επιτροπή, θα ήθελα στην δευτερολογία σας να μας μιλήσετε περισσότερο για την πολιτική βούληση της Επιτροπής να απλοποιήσει τη, τις διαδικασίες. Εγώ προέρχομαι από το, την περιοχή του, στο κέντρο της Γαλλίας και γνωρίζω το πρόβλημα που, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αγρότες μας. Ε, πρέπει να συμπληρώσουν εξαιρετικά περίπλοκες αιτήσει μέσω ίντερνετ και στο τέλος δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να λάβουν ως επιδότηση. Ε, είναι ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να απλοποιηθεί και για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων από την πλευρά της διοίκησης. Και τέλος, στο πλαίσιο στο, του προγράμματος ε, δράσης μας, ίσως θα έπρεπε να ε, προγράμματος εργασιών μας, να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί κύριε Επίτροπε συζητούμε τώρα για διορθώσεις που έγιναν ε, κατά τη διάρκεια πολλών ετών εναντί κρατών μελών Μήπως θα χρειαζόταν μια διαδικασία απαλλαγής πολυετή, δηλαδή που να καλύπτει πολλά χρόνια, πολλά έτη, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται και καλύτερα ο πολίτης. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το διάστημα εμπιστοσύνη σημαίνει ότι το 95% των ε, επιδοτήσεων ε, δίδεται καλώς και το 5% έχει πρόβλημα. Αναρωτιέμαι αν ε, έτσι πρέπει να διαβάσω αυτό το ποσοστό. Συμπερασματικά σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Από ό,τι κατάλαβα στην επόμενη θητεία σας θα σας υποστηρίξει η Ίγκια και η Γερμανία. Από την πλευρά της Γαλλίας μάλλον δεν θα λάβω θέση ακόμα. Θέλω να δω τι θα γίνει και με το ποσοστό τις δημοσιονομικές διορθώσεις έναντι της Γαλλίας πριν να πάρω θέση. Και δεν θέλω να σας συγκρίνω με τον προκάτοχό σας, αλλά συγχαρητήρια για το έργο που επιτελέσατε. Ευχαριστώ. Κύριε Οντή. Ε, γοητευτικοί οι Γάλλοι όταν μιλούν έτσι. Ε, Γιάννης Γκάιερ, έχει το λόγο, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους να ευχαριστήσω και εγώ το ελεγκτικό συνέδριο, τον Επίτροπο, είναι αυτό που μας είπε. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω αν αισθάνεστε σαν ε, ένα χαμστεράκι στο, στον κύκλο του. Στο, δηλαδή τρέχετε, τρέχετε για να μείνετε στο ίδιο σημείο. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ξέρετε πως η δικιά μας πολιτική οικογένεια ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη με τις προτάσεις σας για μεταρρυθμίσεις γεωρικής ε, πολιτικής και υποστηρίξαμε αυτά τα οποία ε, προτείνατε. Αλλά βεβαίως ε, πρέπει να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ήταν αυτό το οποίο στένισε πάρα πολλές από τις καλές σας προτάσεις. Και σβήνει το μικρόφωνο του μελτή. Οπότε αυτό προσπαθούσα να πω με την ερωμίωσή μου ότι σας ε, καθιστούμε υπεύθυνο για πράγματα τα οποία ε, εμείς οι ίδιοι δεν κάναμε. Τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ πέρα πως ακριβώς ε, έχουμε τον τομέα με τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί όπου ακριβώς εμφανίζονται τα περισσότερα προβλήματα και λογικό είναι να μας ανησυχεί περισσότερο. Βεβαίως ε, πάντα έχουμε αυτό το πρόβλημα με την Κομισιόν, το πώς θα γίνουν οι δημοσιονομικές διορθώσεις πιο αποτελεσματικές στη στιγμή που χάνονται λεφτά για τα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά 1,2 δισεκατομμύρια είναι ένα πάρα πολύ ε, εντυπωσιακό νούμερο, αλλά βεβαίως ο χρόνος που χρειάζεται μας προβληματίζει. Εδώ πέρα πρέπει να συμφωνήσω με την κυρία Γκρέσλε. Δηλαδή ε, όλοι αυτοί οι μακροσκελείς ε, διαδικασία φαίνεται πως ε, καθιστά και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα πολύ ασθενέστερο. Τώρα, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Κομισιόν είναι σαφώς γρηγορότερη. Έχει νόημα να εναρμονίσετε τις διαδικασίες μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Δηλαδή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας μήπως θα μπορούσε να δανειστεί τεχνογνωσία από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία από ό,τι φαίνεται ε, εφαρμόζει κάποια πολιτική με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δεύτερο ερώτημα. Χτες είχαμε όχι μια διαφωνία, θα έλεγα μια διαφορά στην εκτίμηση με τον Επίτροπο Χάν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ περήφανος για το ότι πόσο 10-12% των ε, υπαλλήλων του ε, απασχολείται στον έλεγχο. Ήταν περήφανος. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσοι δικοί σας υπάλληλοι απασχολούνται στον έλεγχο και πως θα επιταχύνονταν οι διαδικασίες εάν ε, ε, ακόμη περισσότεροι έκαναν αυτή τη δουλειά. Και τελευταίο ερώτημα. Ένα ερώτημα με το οποίο θα προσπαθήσω πάλι να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Εάν ε, πράγματι με τη βοήθειά μας επιταχυνθούν διαδικασίες, ε, πόσο γρήγορα αναμένετε εσείς αποτελέσματα και αποτελέσματα εννοώ μειωμένο ποσοστό σφάλματος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Ο κύριος Μίλντερ κατόπιν. Ευχαριστώ. Για πολλά χρόνια ο πρώτος πυλώνης ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία ελέγχου του προπολογισμού, γιατί το, το ποσοστό σφάλματος ήταν κάτω του 2%. Πέρυσι όμως άλλαξαν τα πράγματα και όλοι εκπλαγήκαμε. Γιατί όλοι έλεγαν ότι το ΩΣΔΕ είναι ένα εξαιρετικό σύστημα, εξαιρετικά απλό και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι εύκολο να γίνει ο έλεγχο, θα έπρεπε να είναι εύκολο να γίνει και η διόρθωση. Ωστόσο, το ποσοστό σφάλματο που ερχόμαστε να ε, δούμε μπροστά μα ε, φέτο είναι ακόμα υψηλότερο. Και ποια είναι η εξήγηση ότι οι μόνιμοι ε, χορτολιβαδικέ εκτάσει δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά Εάν αυτό ήταν το πρόβλημα και αφού είχαμε στη διάθεσή μας το ΩΣΔΕ, γιατί δεν κατάφερε η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το θέμα νωρί και να επιστρέψουμε στα παλαιότερα ποσοστά του 2% και τα μικρότερα. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, έχουμε πολλές, ε, πολλά ερωτήματα και πολλές παρατηρήσεις εύστοχες από τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε τις απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Πίπερ. Ε, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις στις οποίες είχα ήδη απαντήσει στην ε, παρέμβασή μου, στην πρωτολογία μου, αλλά θα επανέλθω. Μιλήσατε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κράτη-μέλη, για προβλήματα τα οποία είχαν επισημανθεί το 2007, 2008 και παραμένουν το 2013 και πράγματι το διάστημα είναι μεγάλο. Όμως επ' αυτού θα ήθελα να επιμείνω στο εξής. Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν διεξάγει ελέγχους και αναλύσεις είναι να εξασφαλίσει επαρκώς την σωστή και ορθή χρήση των ε, ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και αν θεωρήσει ότι αυτό δεν, έχει, δεν ισχύει, ε, προβαίνει σε διορθώσεις. Το σύστημα αυτό λειτουργεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ε, εκτείνεται στη διάρκεια πολλών ετών, που σημαίνει ότι αν εντοπιστεί σήμερα ένα πρόβλημα, μπορούμε να γυρίσουμε 24 μήνες πίσω στο χρόνο και να ε, ελέγξουμε την κατάσταση. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Τώρα, μπορεί να αντιμετωπίσουμε σήμερα ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, το οποίο να υφίστατο και πριν δύο χρόνια. Έτσι λοιπόν, εάν συμβεί αυτό, επιβάλλουμε δημοσιονομικές διορθώσεις και το εν λόγω κράτους μέλος παραμένει υπό μια κατάσταση παρακολούθησης, παρακολουθεί επί ένα ή δύο χρόνια μέχρι να βεβαιωθούμε ότι ε, το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Χρειάζεται λοιπόν επαρκές χρονικό διάστημα για να μελετήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης στα κράτη-μέλη και υπάρχουν και ιδιαιτερότητες από, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ο Γενικός Διευθυντής ε, πρέπει να υποβάλει μια έκθεση ετήσια η οποία καλύπτει την κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός ε, έτους. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε ότι όταν το ποσοστό σφάλματος είναι κάτω του 2%, ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα να θέσει ε, επιφύλαξη σε σχέση με τη διαχείριση ενός κράτους μέλους. Αυτό είναι αντικειμενικό, δεν μπορούμε να βασιστούμε στην φήμη, στο παρελθόν ενός κράτους μέλους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να εκφραστεί μια επιφύλαξη συστημική όσον αφορά μια γενικότερη αξιολόγηση του πώς λειτουργεί η κατάσταση σε ένα κράτος μέλος. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, μάλλον το, συνολικό ποσοστό σφάλματο δεν ξεπερνούσε το 2% και γι' αυτό ο γενικό διευθυντή δεν εξέφραζε γενική οικονομική επιφύλαξη. Προβλέπαμε όμως ότι το ποσοστό θα ξεπεράσει το 2%. Το βλέπαμε στις αναλύσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο έχει βελτιώσει τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ποσοστού σφάλματος, χρησιμοποιώντας και νέα ε, στοιχεία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, με τον, με τον Γενικό Διευθυντή, καταγράψαμε μια επιφύλαξη οικονομικού ε, χαρακτήρα, δημοσιονομικού χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά έχουμε τις αιτήσεις εκθέσεις. Στις αιτήσεις εκθέσεις αυτή τη στιγμή το ποσοστό σφάλματος του συνολικό ξεπερνά το 2%. Ο Γενικός Διευθυντής καταγράφει ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν υψηλό ποσοστό σφάλματος, το υψηλότερο, και υπολογίζει. Εάν ε, είχαμε, δεν είχαμε συνυπολογίσει το, το ποσοστό σφάλματος για τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Γαλλία, το μέσο ποσοστό ασφάλματος θα ήταν κάτω του 2%. Γι' αυτόν τον λόγο, εξαιτίας αυτών των τριών κρατών μελών, ε, εισήχθη η δημοσιονομική επιφύλαξη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η δημοσιονομική επιφύλαξη εφαρμόζεται μόνο στα τρία κράτη-μέλη, εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε λάβει μέτρα έναντι όλων των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά, αυτή η προσπάθεια διόρθωσης της κατάστασης στα κράτη-μέλη συνεχίζεται μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει βεβαιωθεί. Αυτό συνέβη για την Πορτογαλία, για την ε, Βουλγαρία, για την Ρουμανία. Η Ρουμανία δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στην ε, δημοσιονομική επιφύλαξη γιατί έχει ήδη πληρώσει τη δημοσιονομική διόρθωση. Για αυτές τις τρεις χώρες λοιπόν μαζί και με την Πορτογαλία, μιας και υπήρχε η γενικότερη συστημική επιφύλαξη προηγούμενη και είχαν ε, δημιουργηθεί σχεδιαδράσεις, δημιουργήθηκαν σχεδιαδράσεις τα οποία άρχισαν να υλοποιούνται και μάλιστα στην Πορτογαλία μετά από αυτή την ε, εφαρμογή του σχεδίου δράσης οι δύο τελευταίοι ε, έλεγχοι διαπίστωσαν ότι η κατάσταση έχει διορθωθεί. Παρ' όλα αυτά, ο Γενικό Διευθυντή στην περίπτωση τη Πορτογαλία θέλει να κάνει και ένα δεύτερο έλεγχο για να βεβαιωθεί 100% ότι ε, τα προβλήματα διορθώθηκαν και το ΩΣΔΕ αξιοποιείται. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός, η διαδικασία όλη αυτή μας αναγκάζει να ε, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να εξετάσουμε και να επιλέξουμε τα προβλήματα. Το 2011 μπορούμε να επισημάνουμε και να επιβάλλουμε διορθώσεις για προβλήματα ε, από το 2009 και μετά, για παράδειγμα. Τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται από αυτό το σύστημα ε, καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεύτερον, έχετε δίκιο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας δεν ήταν επαρκή για να ενθαρρύνουμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να επιλύουν τις, ε, τα προβλήματα. Γιατί αυτό, γιατί η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων παίρνει χρόνο. Δεν μπορούν όλα να γίνουν αυτοματοποιημένα. Υπάρχουν και νομικές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το δικαίωμα ε, κατά την παράσταση ε, εξέτασης του κράτους μέλους. Έχει το δικαίωμα το κράτους μέλος να αντιταχθεί στην απόφαση της Επιτροπής να υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι ο τρόπος υπολογισμού της νομοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή δεν είναι σωστός και να αποδείξει ότι το ποσοστό σφάλματος είναι μικρότερο. Είναι η διαδικασία ε, της ε, συνδιαλλαγής. Εξετάζουμε αν μπορούμε κάποια από αυτά τα βήματα αυτής της διαδικασίας να συμπτυχθούν έτσι ώστε να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα, να μην χρειάζονται χρόνια μετά την διαπίστωση του προβλήματος. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε και άλλα κίνητρα προς τα κράτη-μέλη, όχι μόνο την επιβολή της δημοσιονομικής διόρθωσης, της οποίας ο προστασιακός στόχος είναι η προστασία των οικονομικών σφαιρών της Ένωσης, αλλά επίσης και άλλα κίνητρα, όπως εκείνα που εισήχθησαν με τον νέα ΚΑΠ, δηλαδή το... η δυνατότητα διακοπής των επιδοτήσεων. Υπήρχε αυτή η διαδικασία και παλαιότερα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και καθόλου αποτελεσματική. Με τον νέο κανονισμό θα έχουμε αυτή τη ε, δυνατότητα στα χέρια μας. στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης έχουμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε τέτοιες ε, διακοπές ε, των επιδοτήσεων. Από το 2014 και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε αυτό και στον δεύτερο πυλώνα και στην και στο, στο, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στον πρώτο πυλώνα δεν έχει και πολύ νόημα γιατί πρόκειται για άμεσες επιδοτήσεις. Αλλά αυτές, αυτός ο μηχανισμός θα είναι επίσης ένα κίνητρο για τα κράτη-μέλη να ε, διορθώνουν τα προβλήματα. Έγιναν ε, μεγάλες αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Και γι' αυτό, όπως είπε ο κ. Γκάιερ, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εισήχθησαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα τα επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους απλοποίησης. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν, ε, παραμένει μια απλοποίηση των διαδικασιών στον δεύτερο πυλώνα, οι απλοποιημένες ε, ε, πληρωμές, οι καταποκοπήν υπολογισμοί, στα προγράμματα που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη θα συμπεριλάβουμε και κριτήρια ε, για την, ε, τον, έλεγχο, τον επιτόπιο έλεγχο καθώς επίσης και για, τους, για τον τρόπο μάλλον με τον ορισμό των επιλέξιμων περιοχών και των μόνιμων χορτοβολ... λιβαδικών εκτάσεων έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε καλύτερα την, υπόψη μας την κατάσταση ε, επιτόπου. Από τη στιγμή που ελήφθη η, απόφαση για την αποσύνδεση, λαμβάνουμε υπόψη μας στον ορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων την πραγματική κατάσταση των αγροτεμαχίων. Γιατί διαφορετικά είχαμε ε, πιο περίπλοκες διαδικασίες που δεν είχαν νόημα. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία απλοποίησης. Αυτή η απλοποίηση σε συνδυασμό με τα κίνητρα που εισήχθησαν στην νομοθεσία νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος. Με το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και με το σύστημα καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. 1 δισεκατομμύριο ευρώ αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των ε, χρηματοδοτήσεων για την ΚΑΠ. Αυτό ήταν το ποσοστό σφάλματος έω τώρα. Διαπιστώνεται ότι αυξάνεται το ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων και αυτό επειδή το σύστημα λειτουργεί, επειδή εντοπίζονται τα προβλήματα. Και όταν εισπράττονται αυτές οι δημοσιονομικές διορθώσεις προστατεύονται τα συμφέροντα του προπολογισμού της Ένωσης, αλλά επίσης πρέπει να διορθωθεί και η γενικότερη κατάσταση. Ο μηχανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη προστατεύει τα συμφέροντα της, Επιτρο... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχων οι οργανισμοί πιστοποίησης αναλαμβάνουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο και χρειάστηκε να ε, ε, προσαρμόσουμε και εμείς τον τρόπο ελέγχου έτσι ώστε να συνεργαζόμαστε πιο στενά με αυτούς τους οργανισμούς πιστοποίησης. Ε, επομένως συνεργαζόμαστε με αυτούς στον τομέα της πιστοποίησης, της τεχνικής βοήθειας, Πολλά μέτρα πρέπει να ληφθούν από εδώ και πέρα νωρίτερα και νομίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους ενίσχυσης της ευθύνης των κρατών μελών. Γιατί όπως διευκρίνησε το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι λάθη τα οποία έχουν βρεθεί θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί από τα κράτη-μέλη πλασιάσαμε το προσωπικό ελέγχων, ε, έχουμε μια διεύθυνση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας που ασχολείται με θέματα ε, τέτοιου ελέγχου, αλλά δεν ε, επιμένουμε αποκλειστικά στις, σε εισαγωγικά τιμωρητικές αν θέλετε δράσεις, θέλουμε να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με νωρίτερες παρεμβάσεις οι οποίες θα λαμβάνονται νωρίτερα και θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες πληρωμών έτσι ώστε να λειτουργήσουν με συστούς ελέγχους και με διαδικασίες ελεγκτικές απλούστερες. Όπως διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο, πολλά προβλήματα δημιουργούνται γιατί οι εθνικές διαδικασίες είναι περίπλοκες και άλλα καταλαβαίνουν οι ελεγκτές, άλλα αυτοί οι οποίοι καλούνται να ωφεληθούν από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Για την κυρία Γκρέσλε να ε, είχε θέσει κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις εν μέρη μόνο απάντησα πως ε, ε, το ποσοστό αυτό λάθος το τελικό υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε δεν επαφιέμεθα στις διαβεβαιώσεις των γενικών διευθυντών των μηχανισμών πληρων, των υπηρεσιών πληρωμών αλλά ε, έχουμε δημιουργήσει νέους δείκτες ποιοτικούς που λαμβάνουν υπόψη φυσικά τους ελέγχους που έχουν γίνει από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας αλλά και τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία γίνονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Όλοι αυτοί οι δείκτες ε, ομαδοποιούνται και μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το ποσοστό σφάλματος το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το σύστημα αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από το δημοσιονομικό έτος 2014 υπευθυνοποιώντα και τους μηχανισμούς πιστοποίησης που θα πρέπει να ξανακάνουν ένα αντιπροσωπευτικό δειγματολόγιο σε κάθε κράτος μέλος που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα και αν διπλασιάσουμε εκ νέου τον αριθμό των ελεγκτών οι οργανισμοί πιστοποίησης θα το κάνουν αυτό και θα συνεργαστούμε μαζί τους για να τις βοηθήσουμε, για να τους βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Είχα εξηγήσει γιατί υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των διαφόρων κρατών μελών και γιατί υπάρχουν ε, <clears throat> δημοσιονομικές ε, ε, διορθώσεις διαφορετικές με τις ετήσιες εκθέσεις επιβάλλεται αυτή η διόρθωση ανεξάρτητα αν υπάρχει αποθεματικό μόνο και μόνο γιατί διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα. Γιατί αυτό απαιτεί η προστασία του προϋπολογισμού. Από την άλλη όμως η ετήσια έκθεση που είναι μια φωτογραφία αν θέλετε την οποία κάνουν σε ετήσια βάση βέβαια οι γενικοί διευθυντής δημιουργούν κάποιες, κάποιες προβλέψεις ε, ακόμα και αν το ποσοστό δεν ξεπερνά το 2%. Δημιουργούν ένα είδος αποθεματικού ακόμα και αν το ποσοστό σφάλματος δεν περνά το 2%. Αναφερθήκατε στην ελληνική υπηρεσία. Η Ελλάδα ε, για πολλά χρόνια υπέστη τέτοιες διορθώσεις και έχει αρχίσει να επιστρέφει τώρα γιατί τερματίζεται όπως είπα το μορατόριο, γιατί το πρόγραμμα δράσης δεν τέθηκε απολύτως σε λειτουργία εν μέρη μόνο και γι' αυτό διεκόπη το μορατόριο και ζητήσαμε, αρχίσαμε να ζητάμε επιστροφές. Όμως το σύστημα LPIF έχει στην ουσία ξανασχεδιαθεί από την Ελλάδα, ε, έχει πληρώσει λοιπόν ε, η Ελλάδα όχι μόνο τις διορθώσεις αλλά και το νέο σύστημα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε περισσότερες διαβεβαιώσεις σχετικά με την ποιότητα της βάσης δεδομένων. Τώρα το θέμα του ελέγχου τίθεται. Το θέμα είναι πώς οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τη βάση αυτή δεδομένων και τι λάθη μπορεί να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ο οργανισμός ο οποίος θα μας δώσει την διαβεβαίωση για την Ελλάδα δεν θα είναι η υπηρεσία πληρωμών αλλά ο μηχανισμός πιστοποίησης, ο οργανισμός πιστοποίησης που είναι κάτι το διαφορετικό και ανεξάρτητο από την υπηρεσία πληρωμών. Άλλη ερώτηση. Η αλλαγή της μεθοδολογίας του συνεδρίου. Πέρυσι συζητήσαμε ε, κατά πολύ με το συνέδριο τα θέματα της μεθοδολογίας. Το είχα πει και πέρυσι ότι εγώ δεν θα σχολιάσω τη μεθοδολογία της και έχει δικαίωμα να την επιλέγει το συνέδριο. Εμείς θεωρούμε πάντως όταν έχουμε διαφορετική άποψη ότι πρέπει να πούμε τη γνώμη μας. Ε, είχα πει σαν παράδειγμα η οικοαιρεσιμότητα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι δεν έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί γιατί αυτή η οικοαιρεσιμότητα δεν είναι κριτήριο επιλεξιμότητας για να περάσει κανείς σε άμεσες πληρωμές. Όμως το ότι δημιουργήθηκε αυτό το, ε, αυτή η προϋπόθεση φτάνει το 0,2% για τον πρώτο πυλώνα. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλες διαφωνίες με το ε, συνέδριο το ελεγκτικό για το μεσοδιάστημα τώρα μέσα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και να μετρηθεί ένα ποσοστό σφάλματος ε, χρειάστηκε να βελτιώσουμε εμείς το σύστημα υπολογισμού αυτού του ποσοστού σφάλματος ορίζοντας καλύτερα το λεγόμενο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Για τον κύριο Οντί αναφερθήκατε στο θέμα του δειγματολογίου του συνεδρίου και εδώ θα πρέπει να απαντήσει το συνέδριο και όχι εγώ για τις ειδικέ εκθέσεις για το πώς έχουν δαπανηθεί τα χρήματα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς αυτό κάνουμε ή τουλάχιστον αυτό θεωρούμε ότι κάνουμε. Από τη μία προσπιζόμεθα τα οικονομικά συμφέροντα και από την άλλη ο Επίτροπος είναι υπεύθυνο για τα σωστά αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς υπεύθυνοι μόνο για τη σωστή χρήση των πιστώσεων, αλλά και την δημιουργία ε, των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Αν θέλουμε εμείς ε, να αφαιρέσουμε από την ανάπτυξη της υπαίθρου ό,τι περιπλέκει τα πράγματα, τότε θα μείνουμε μόνο με τρία-τέσσερα μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται με καθολικό και ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις πολιτικές απαιτήσει και τους στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε εδώ μια επιλογή. Θέλουμε εμείς ένα μαθηματικά χαμηλό, πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματος χωρίς πολιτικούς στόχους ή μήπως θέλουμε να έχουμε και πολιτικούς στόχους οι οποίοι να εφαρμόζονται με μέτρα τα οποία θα μας επιτρέξουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ελεγξιμότητας. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε. για την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις περιφέρειες και τη γενική μας διεύθυνση. Γίνεται αυτή η προσπάθεια συντονισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις γενικές διευθύνσεις οι οποίες είναι σε σύστημα κοινή διαχείρισης. Και έχουμε και τον λεγόμενο οριζόντιο κανόνα που καλύπτει όλες τις γενικές διευθύνσεις. Για τις ανακτήσεις ποσών όμως και τις ε, διακοπές και τις διορθώσεις, συγγνώμη, ε, για τη γεωργία ε, ήταν καθαρές οι διορθώσεις αυτές, οπότε αυτό το οποίο παίρνουμε πίσω σαν χρήματα και τα οποία ξαναγυρνούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγαιναν απευθεία στον προϋπολογισμό της Ένωσης και όχι πλέον στα κράτη-μέλη. Τώρα η διαδικασία εναρμονισμού από το 2014 θα συνεχιστεί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη. Για τον κύριο Μίλντερ, για το ΙΑΞ. Και εγώ είπα στην εισαγωγή μου ότι εξακολουθώ να θεωρώ ότι το σύστημα αυτό ως δε ως έχει είναι ένα καλό σύστημα σε σχέση με το σύστημα πληρωμών που έχουμε ε, με την επιφάνεια, για ε, την επιφάνεια. Γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα μέχρι τώρα και ξαφνικά τώρα δημιουργήθηκαν προβλήματα. Αυτό είναι καρπός της ανάλυσης την οποία συνέλεξα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εδώ και αρκετό καιρό, θα δείτε ότι αν δείτε τι έγινε το 2002, 2003 και 2004 και δείτε τους ελέγχους που είχαν γίνει επιτόπια, θα δείτε ότι βασιζόντουσαν σε ένα συνδεδεμένο με την παραγωγή σύστημα. Υπήρχε μια πληρωμή δηλαδή για τις επιφάνειες οι οποίες είχαν συγκεκριμένους τύπους παραγωγής. Ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος ο ορισμός τους λοιπόν και ο κίνδυνος λάθους και για αυτούς οι οποίοι έπαιρναν τα χρήματα και για τους ελεγκτές ήταν μικρός. Αν ένα, μια γεωργική επιφάνεια είχε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια ήταν επιλέξιμη. Από το 2005 και μετά υπήρξε η αποσύνδεση και αυτό φάνηκε κυρίως μετά το 2006-2007, λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή, γιατί αυξήθηκε για πληρωμές η επιφάνεια η οποία ήταν επιλέξιμη ε, και η οποία απλά έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλέξιμη. Οπότε τότε ε, ε, αυξήθηκε ο αριθμός των γεών δυνητικά καλλιεργήσιμων ακόμα και χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί βέβαια με εντατικό τρόπο. Και εκεί ξεκίνησαν προβλήματα και σε σχέση με την ποιότητα των συγκεκριμένων εκτάσεων και σε σχέση με τους ελέγχους τους επιτόπιους. Εμείς παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν από το 2014 γιατί ήδη στην παρούσα μεταρρύθμιση έχουμε επανεξετάσει το θέμα των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων όπως επίσης και των επιλέξιμων επιφανειών για να μην είμαστε δίσκαμπτοι στον τρόπο ορισμού και χαρακτηρισμού των γεών. Γι' αυτό συνεχίζω να πιστεύω ότι το σύστημα ως έχει δεν είναι κακό, αλλά θα πρέπει εμείς να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, όπως επίσης και μια ολόκληρη σειρά παρεμβάσεων για την αύξηση της ποιότητας του ελέγχου και της ποιότητας φυσικά των ελεγκτών. Σα äh, Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Βλέπετε γιατί οι είναι άμεσες ο κύριος Πίπερ. Πρώτος και μετά η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Πρέπει να αναγνωρίσω πως οι απαντήσεις που δώσατε είναι πίστικες και προσέφεραν και κάποια επιπρόσθετα πράγματα κυρίως το ότι τα λάθη τα οποία βρίσκεται απλά έχουν γίνει στο παρελθόν, γι' αυτό φαίνεται ότι τραβάνε τόσο πολύ οι διαδικασίες. Αυτό μου φαίνεται λογικό πράγματι. Παρ' όλα αυτά, έχω σοβαρά προβλήματα ε, με αυτό το οποίο προβλέπεται για το μέλλον, το εάν θα συμβεί κιόλας. Είναι σαφές όταν μιλάμε για απλοποίηση της γεωργικής ανάπτυξης ε, πως ε, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω με κάποια λύση κατά θα μπορέσει να πέσει το ποσοστό σφάλματος ε, το 6,8% νομίζω σε σύγκριση με άλλες πολιτικές είναι πάρα πολύ ψηλό και το εάν θα γίνει όντως ε, αυτό το οποίο λέτε. Θα το δούμε, αν γίνει θα μας χαροποιήσει. Ε, τώρα, αυτό το οποίο βεβαίως δεν μας διαφωτίζει είναι αυτά τα οποία μας είπατε για το σύστημα των εκτάσεων. Εγώ πήγα με το αυτοκίνητο στην Πορτογαλία σε περιοχές της Υπέθρου της Γερμανίας ε, άνοιξα το GPS για να αποφύγω ένα μποτιλιάρισμα και βρε... βρέθηκα σε κάτι χωράφια. Έτσι και βλέπω εκεί πέρα σε ένα απλό GPS που βρίσκομαι, έτσι, χωρίς να οδηγάω καμιά λιμουζίνα. Όταν υπάρχουν και συστήματα όπως το Google Earth, νομίζω θα μπορούσαμε να βρούμε το που είμαστε. Ε, εγώ με το GPS βρήκα τα πάντα. και δεν μπορώ να καταλάβω πως σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία ή η Γαλλία από το 2007 υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Έπρεπε να έχει συμβεί κάτι και αναμένουμε πολύ γρήγορα να συμβεί κάτι. Όσον αφορά τις ε, καθαρές ε, διορθώσεις, ε, ήσταν κάπως αφήσει, Είπατε πώς θέλουμε να περιορίσουμε τις διαδικασίες από τα 5 στα 2 έτη. Αλλά συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό. Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα. Αυτές τις ερωτήσεις έχω εγώ. Να ακούσουμε και την κυρία Γκρέσλε. Παρακαλώ. από το Σαββατοκύριακο παλεύω με όλα αυτά τα χαρτιά εδώ πέρα. Έχω την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Γενικού Διευθυντή, τις ανακοινώσεις για τις διορθώσεις και προσπαθώ να, να τις καταλάβω. Να αφαιρθώ στο Ελπίες. Είναι πρόβλημα σε πολλές χώρες, το ανέφερε και ο κύριος Πίπερ, στην, Πορτογαλία είναι γνωστό από το 2006. Η Κομισιόν έχει και μία επιφύλαξη. Στη Βουλγαρία 2008, στη Γαλλία από το 2007. Έκτοτε δηλώνουν αυτέ οι χώρες ε, κάποιες εκτάσεις ε, ως ε, μόνιμες καλλιέργειες χωρίς να είναι... Μα αυτά ε, δεν μπορεί να είναι λάθη έτσι. Μήπως υπάρχουν χώρες οι οποίες το κάνουν και εμένα. Το γιατί θα κάνουν κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο κέρδος από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δούμε τις διορθώσεις, αν δούμε τα ποσά των ε, διορθώσεων, είναι σε τελική ανάλυση γελία. Δηλαδή οι κυρώσεις σε σύγκριση με το κέρδος δεν είναι τίποτα. Ε, εκεί είναι το πρόβλημα. Λέω συνέχεια πως δεν θέλω τα λεφτά, αλλά θέλω να αλλάξει το, το σύστημα. Αλλά το ερώτημα είναι τελικά. Από πότε η Κομισιόν είναι ενήμερη για αυτό το πρόβλημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι συστημικό. Και ε, αυτό το οποίο λέτε δημοσιονομική διόρθωση ε, είναι γελία, έτσι. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποια κράτη-μέλη επηρεάζει αυτό το πρόβλημα και πόσο ε, εκτιμάτε εσείς ότι είναι οι συνέπειες αυτού του προβλήματος. Εγώ θεωρώ πως είναι πλέον κάτι εσκεμμένο, δεν είναι σφάλμα και αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο για την Ελλάδα. Έχω πάει και δύο φορές με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και με συγχωρείτε ε, οι συνάδελφοι από την Ελλάδα, αλλά είπατε εντάξει μορατόριο σταμάτησε, αλλά μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ που ξανά ε, έλεγαν τον Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, είχα πάει και το 2007 και το 2010 στην Ελλάδα και κάθε φορά ορκιζόταν η Κομισιόν πως λειτουργεί το σύστημα. Ε, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί όμως. Αν μετά από τρία χρόνια μας λέτε ε, πως τώρα λειτουργεί αλλά τις προηγούμενες φορές δεν λειτουργούσε, ε, κάποιος μας δούλευε δηλαδή. Λέτε πως το πρόβλημα το ξέρουμε το 2006 και δεν έχει λυθεί ακόμα. Από το 97 ήδη όταν είχε ξεκινήσει το ΩΣΔΕ. Τώρα λέτε πως αποτελέσματα θα έχουμε το 2015. 15. Γιατί, γιατί τότε εξακολουθείτε να δίνετε λεφτά. Μάλιστα. Jean-Pierre Ευχαριστώ τροφή προ συζήτηση. Για σκέψη μάλλον. Σε σχέση με αυτό που είπε και η Βλέπουμε ότι η κοινή διαχείριση έχει πλέον κλείσει τον κύκλο της. Κύκλο της. Παλαιότερα ε, κάτι εξυπηρετούσε, αλλά πλέον δεν έχει νόημα. Ίσως πρέπει να κάνουμε μια μελέτη τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα έπρεπε να κάνει μια μελέτη να την αξιολογήσει. Κύριε Επίτροπε, λέτε ότι θα κάνουμε συνοδευτικούς ελεγχούς βασιζόμενοι και συνεργαζόμενοι με τους οργανισμούς πιστοποίησης. Ναι, μια χαρά, αλλά όταν εδώ με τη συνάδελφο είχαμε πάει στη Γαλλία για να εξετάσουμε την κατάσταση σε μια ε, τέτοια εποπτεύουσα ε, αρχή, οργανισμό πιστοποίησης μάλλον, μου δημιουργήθηκε εντύπωση, μάλλον αντιλήφθηκα, ότι δεν ήταν ανεξάρτητη, γιατί υπάγονταν κάτω από το Υπουργείο. Δεν θα έπρεπε ε, να το ξανασκεφτεί αυτό το ζήτημα η Επιτροπή. Γιατί τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση για να ε, ασκούν αυτούς τους ελέγχους. Εκεί πρόκειται για πραγματικά ανεξάρτητους ελεγκτές και όχι για δημόσιους υπάλληλους ε, των κρατών μελών. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι την κοινή διαχείριση θα έπρεπε να την καταργήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού την κρατάμε, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα ασκούμε τον έλεγχο στην κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ πλήρω με την γκια σε αυτά. Σα ευχαριστώ. Ξεχάσατε κάτι κυρία Γκρέσλε. Ναι, κύριε Επίτροπε για τη Ρουμανία. Έχουμε σοβαρή αλλαγή του ποινικού δικαίου. Είναι πλέον ε, ε, και για ποινικά δικήματα μη υπόλογη η πολιτική. Ε, πώς το εκτιμάτε αυτό. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα και εγώ να κάνω μία κύριε Επίτροπε. από αυτά τα οποία είπατε και από τις ερωτήσεις των βουλευτών υπάρχει εντύπωση πως ε, υπάρχει ένα πρόβλημα ελέγχου των κονδυλίων που είναι το ότι έχουμε πολύ περίπλοκη νομοθεσία. Υπάρχει δηλαδή μια σχεδιασμένη οικονομία ε, ως προσέγγιση Πώς το βλέπετε, εσείς μιλάτε για βελτιώσεις που θα γίνουν. Τώρα έχουμε μια νέα γεωργική πολιτική που εγκρίθηκε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, θα γίνει απλούστερη κατάσταση με τη νέα νομοθεσία ή δυσκολότερη. Euh, Για τον κύριο Πίπερ. Για τον δεύτερο πυλώνα. Πώς να μειώσει κανείς το ποσοστό σφάλματος. Εγώ το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Σας το είπα και πέρυσι. Εάν πράγματι θέλουμε να κρατήσουμε μια πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου με στόχους ικανούς να βοηθήσουν τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε ένα ποσοστό λάθους κάτω του 2% με το σημερινό σύστημα υπολογισμού του λάθους. Γι' αυτό είχα διανύμει και ένα κατάλογο με παραδείγματα χρηστών πρακτικών και προγραμμάτων που ε, μπορεί να ισχύουν κυρίως σε θέματα δημοσίων προμηθειών ότι είναι λάθος 100% αλλά ο βασικός στόχος επιτυγχάνεται. Λοιπόν, αν στόχος είναι να πέσουμε κάτω από το 2% θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως το ποσοστό λάθος θα πρέπει να μειωθεί και με αυτή την επιφύλαξη. Γιατί το 7% με αυτή την επιφύλαξη είναι ψηλό. Πρέπει να μειωθεί. Το πώς θα γίνει Είχα ήδη δώσει κάποια παραδείγματα οριζόντιων μέτρων τα οποία καλούμαθα να πάρουμε για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να είναι πιο προσεκτικά σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων γιατί το ελεγκτικό συνέδριο παρατήρησε ότι τα προβλήματα πολλές φορές μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν σε επίπεδο κράτους μέλους. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να λάβουν τις ευθύνες τους ως συνδιαχειριστές. Και όταν ένα έλεγχος γίνεται από ένα κράτος μέλος πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο. Αλλά υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη στους έλεγκτες και πρέπει εμείς να πάρουμε μέτρα δεσμευτικά για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει όμως ένας βαθμός περιπλοκότητας αντικειμενικής θα έλεγα ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να απλοποιήσουμε κάποιες ρυθμίσεις. Δεν καταστήσαμε υποχρεωτικές ε, για τα κράτη-μέλη κάποιες δηλώσεις σε σχέση με τις καταποκοπήν πληρωμές γιατί ο ορισμός ενός μέτρου ακολουθεί αν θέλετε την επιλογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας από τα κράτη-μέλη και θα ακούσετε ίσως διάφορα κράτη-μέλη και υπουργούς Γεωργίας να διαμαρτύρονται γι' αυτό. Γιατί δεν θα εγκρίνουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου τους, ε, ακόμα και αν είναι σωστή η στόχη, γιατί τα μέτρα που προτείνουν είναι πολλά, πολύ περίπλοκα και δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα κράτη-μέλη τους τρόπους απλούστευσης που έχουμε εμείς θέσει στη διάθεσή τους. Αυτό θα καθυστερήσει την έγκριση ενός προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου. Για τον δεύτερο πυλώνα λοιπόν αυτό μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά μένει να βρούμε τα σωστά προγράμματα και να δούμε αν έχει γίνει σωστά ο έλεγχος και αν δεν έχει γίνει σωστά ο έλεγχος και σας έφερα παραδείγματα για δύο-τρεις χώρες μπορούμε να διακόψουμε τις πληρωμές από τη μία εβδομάδα στην άλλη ότι έτσι λειτουργούν οι επιστροφές τις οποίες ναι. δίνουμε. Και αν τυχόν τα μέτρα δεν είναι ικανοποιητικά διακόπτουμε ε, ε, πλήρως ε, τις πληρωμές. Τώρα για τον πρώτο πυλώνα και για το σύστημα των εκτάσεων. Χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αν και με προκαλέσατε με το GPS του αυτοκινήτου σας κύριε Πίπερ, Υπάρχει ένα επίπεδο διευκρίνησης ε, θα έλεγα διαφορετικό ανάμεσα στο GPS της Google και σε αυτό που ζητάμε εμείς για τον ορισμό των εκτάσεων. Ε, και εγώ έχω κάνει τέτοιες διαπιστώσεις όταν ήμουν υπουργό η Ρωμανία έπρεπε να πληρώσει κάποιες δημοσιονομικές επιστροφές και γι' αυτό κάναμε ελέγχους στις εκτάσεις για να είμαστε σίγουροι για ε, τη συγκεκριμένη οριοθέτηση. Λοιπόν, το επίπεδο ε, λεπτομέρειας είναι διαφορετικό. Το θέμα δεν είναι ο καθορισμός ή ο ορισμός, αν θέλετε, μια έκτασης μέσω του Google. Ε, για τις μεγάλες εκτάσεις, 10 εκταρίων, πολλές φορές ένα τμήμα είναι επιλέξιμο, λόγω των τρόπων που ορίζεται η επιλεξιμότητα των γεών, ε, μέσω των, ε, για τις άμεσες πληρωμές. Γιατί μπορούμε να έχουμε σε ε, μια έκταση σαν παράδειγμα μια μόνιμη χορτολιβαδική έκταση στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Σουηδία κάποια τμήματα που είναι εκτάσεις προς βοσκή και μετά υπάρχουν δάση, μετά υπάρχει ένα άλλο μικρό κομμάτι με χορτολιβαδικές εκτάσεις και μετά πάλι δέντρα και τα κράτη-μέλη αυτό που πρέπει να κάνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς είναι να διαγράψουν αν θέλετε τις περιοχές οι οποίες έχουν δέντρα υψηλά και βράχους. Και εκεί τίθεται το θέμα της ακρίβειας σε πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν με τον ε, κανονισμό που έχουμε τώρα για να αποφύγουμε αυτά τα λάθη γιατί πολλές φορές μια γελάδα ή ένα απρόβατο θα πάει και στα δάση μερικές φορές εφόσον υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί το χόρτο που τα ενδιαφέρει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η χώρα λέει ότι η περιοχή αυτή είναι επιλέξιμη. Ενώ ο ελεγκτής μας ή ο ελεγκτής του ελεγκτικού συνεδρίου λέει όχι δεν είναι επιλέξιμη διότι θα πρέπει να είναι μόνο και αυστηρά χορτολιβαδική. Εκεί λοιπόν υπάρχουν προβλήματα διευκρινίσαμε με πιο σωστό τρόπο το τι σημαίνει ε, μια τέτοια ε, μόνιμη χορτολιβαδική και έτσι μπορέσαμε να διευκρινίσουμε καλύτερα τις ε, εκτάσεις αυτές. Και βάλαμε και ένα περιθώριο 10% για τα κράτη-μέλη όταν ορίζουν τις μόνιμες χορτολιβαδικές να ορίζουν και τις επιφάνειες οι οποίες μπορεί να είναι επιλέξιμες και άλλες να μην είναι. Εκεί υπάρχουν προβλήματα, όχι με τον φυσικό διαχωρισμό και οριοθέτηση των εκτάσεων. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι από το 2014 θα έχουμε μέσα στη διάθεσή μας για να απομακρύνουμε τους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από την λαμφασμένη ερμηνεία του κανονισμού. Διορθώνονται λοιπόν τα προβλήματα. Ε, για την Πορτογαλία ή για άλλα κράτη-μέλη, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα εδώ από το 2007 και μετά. Γιατί από το 2007, από τότε που εντοπίσαμε τα προβλήματα αυτά, αρχίσαμε να τα ρυθμίζουμε, ε, ξανακάνοντας την οριοθέτηση των εκτάσεων χώρα. Αυτό κοστίζει σε κάθε χώρα βέβαια και εμείς δημοσιονομικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε και πρακτικά πολλές φορές να ξανακάνει την εναέρια φωτογράφηση και την ψηφιοποίηση ε, των εκτάσεων όλων μέσα σε ένα χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Όταν λοιπόν ένα κράτος μέλος έχει ένα πρόβλημα με, την, ε, με τις εκτάσεις ζητάμε ε, κάθε χρόνο να παρουσιάζει μια διορθωμένη εικόνα ανά τρίτο κάθε φορά τον χρόνο. Γι' αυτό μια πλήρης αλλαγή απαιτεί τρία ή τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου το κράτος πληρώνει τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η Ελλάδα πλήρωσε το 6% των πληρωμών που ε, πήγαιναν στους γεωργούς, ξαναγύρισαν στον προϋπολογισμό. Βέβαια μπορείτε να μου πείτε ότι το λάθος μπορεί να ξεπερνάει αυτό το 6%. Όμως το συνέδριο παρατήρησε στις επισκέψεις του ότι πολλές φορές οι υπερβάσεις ε, μερικές φορές είναι ελάσσονες. Λίγα μέτρα. Δεν είναι λάθη τα οποία είναι εύκολο να δει κανείς. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα λάθη. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα ε, στην ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη πρέπει ε, βλέπουμε αν θέλουν να κερδίσουν με πλάγιο τρόπο κάτι περισσότερο. Υπάρχει ένας διοικητικός έλεγχος όμως, ο οποίος γίνεται επί τη βάση του χάρτη των εκτάσεων και δεν είναι δυνατό να υπάρξουν απάτες σε μεγάλη κλίμακα. Βέβαια εκεί όπου ο ορισμός ε, της επιλέξιμης ηχής δεν είναι ξεκάθαρος μπορεί να υπάρξει παρερμηνία. Η παρερμηνία αυτή μπορεί να είναι σκόπιμη, μπορεί να είναι θέμα παρανόησης. Για την Ελλάδα το σύστημα έτσι όπως ελέγχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας είδαμε ότι ο χάρτης ξαναφτιάχτηκε από την Ελλάδα και σε επίπεδο βάσης δεδομένων είμαστε, ε, έχουμε ε, την εγγύηση ότι τα πράγματα είναι σωστά. Το θέμα είναι πώς οι ελεγκτές θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη βάση δεδομένων σαν αναφορά όταν κάνουν τους ελέγχους. Αυτό πήρε χρόνο. Τρία χρόνια χρειάστηκαν στην Ελλάδα για να ξαναγίνει ο ορισμός των εκτάσεων και να ψηφιοποιηθεί. Η Ελλάδα βλέπετε λοιπόν ότι έχει έναν προϋπολογισμό πολύ πιο μειωμένο από την Γαλλία ή ε, η διόρθωση δημοσιονομική είναι στο ίδιο ύψος με τη Γαλλία με τα χρήματα που θα πληρώσουν οι Γάλλοι δηλαδή τα ίδια θα πληρώσουν και οι Έλληνες. Και το ίδιο γίνεται και για την Πορτογαλία. Εκεί όπου το πρόβλημα έχει εντοπιστεί ζητήσαμε να ξαναγίνει ε, οριοθέτηση, ξανά αυτό, αλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε κάποια χρόνια. Και στις εκθέσεις τις οποίες διαβάσατε η Πορτογαλία δεν είχε συμπεριληφθεί γιατί δεν υπήρχε επιφύλαξη γιατί στην ουσία το πρόγραμμα δράσης εξελίσσεται από το 2007 μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι σας έχουμε δώσει και ένα πίνακα με τον υπολογισμό των διορθώσεων των δημοσιονομικών που πλήρωσε κάθε κράτος μέλος από το 2007 μέχρι σήμερα και τα προγράμματα δράσης τα οποία ε, συμπεριελήφθηκαν σε αυτά. Τώρα, τα χρήματα τα οποία πήραμε πίσω είναι γελία ένα δις, πάνω από ένα δις. Δεν ξέρω αν είναι γελία, η ποσότητα αυτή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με το ποσοστό λάθος το οποίο έχουμε διαπιστώσει σφαιρικά. Αυτό το ένα δις σε κάποια κράτη-μέλη είναι σημαντικό, αλλά λιγότερο. Θα δείτε ότι ακόμα και μικρές χώρες μερικές φορές πληρώνουν περισσότερα από μεγάλες χώρες αν τα προβλήματα είναι πιο σημαντικά σε αυτές. Ναι, πράγματι η ΚΑΠ είναι 50 δις. Αλλά το ποσοστό λάθος είναι και αυτό σχετικά χαμηλό. Ένα δις στα 50 δις είναι το 2%. Δεν είναι τίποτα. Θα δείτε ότι τα επόμενα χρόνια για τον υπολογισμό των προβλημάτων που εντοπίστηκαν το 2009, 2010 και 2011 οι δημοσιονομικές διορθώσεις θα είναι υψηλότερες. Και υπάρχουν αντιδράσεις από πλευρά ορισμένων κρατών μελών που έχουν αρχίσει τώρα να καταλαβαίνουν ότι κοστίζει αυτό που κάνουν. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος υπουργό που έχει κάνει το λάθος σε εισαγωγικά. Υπάρχει διαφοροποίηση μερικές φορές, αλλά παρόλα αυτά το κράτος μέλος πληρώνει και ότι εμείς θα μειώσουμε ε, την χρονική ε, περίοδο που απαιτείται για να γίνει η διόρθωση είναι και αυτό σημαντικό. Θα μειώσουμε κάποια στάδια ενδιάμεσα στις διαδικασίες. Ήδη κάνουμε κάποιες αναλύσεις, κάνουμε κάποιους υπολογισμούς Έχουμε και την καταντιπαράθεση φάση όπου συζητάμε τα θέματα αυτά από τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη ζητούν χρόνο για να ξανακάνουν δειγματοληψία και να μας δώσουν ένα επακριβέστερο επίπεδο του ποσοστού λάθους. Πολλές φορές δίνουμε τη δυνατότητα αυτή, την ευελιξία αυτή στα κράτη-μέλη για να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Τώρα όμως μειώνουμε ακόμα περισσότερο την περίοδο αυτή και θα συμπτύξουμε ε, κάποια στάδια στις αναλύσεις που κάνουμε για να παίρνουμε πιο γρήγορα τις αποφάσεις και πιο σωστά. Στις εσωτερικές διοικητικές μας δραστηριότητες θα μειώσουμε επίσης τον χρόνο που απαιτείται και θα δώσουμε επίσης ε, την δυνατότητα ενός ελάχιστου χρόνου στα κράτη-μέλη για να υπερασπίσουν τον εαυτό τους χωρίς να, παραμείνουμε, να παρατείνουμε συγγνώμη, τον χρόνο αυτό. Ο κύριος Σοντή έκανε ορισμένες προτάσεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να, τις να συζητηθούν αυτές σε πολιτικό επίπεδο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει ένα μικρότερο περιθώριο ε, ποσοστό σφάλματος, αλλά η ευθύνη βαρύνει ε, και την Επιτροπή και τα κρατη γιατί πρόκειται και κοινή η διαχείριση και τώρα πια δεν είμαστε 15, είμαστε 28. Επομένω, δεν γίνεται να μην εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν ανεξάρτητο οργανισμό σε κράτος ε, μέλος. Γιατί αν αποφασίσουμε ότι δεν εμπιστευόμαστε πλέον τα κράτη-μέλη, τελικά ποιον αποστελεί, ποιος αποτελεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απλώς ένας φορέας, ένας, ε, ένας θεσμός, ένα θεσμικό όργανο με Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί τις πολιτικές που αποφασίζονται στο Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα, δεν μπορεί να μην εμπιστεύεται έναν ανεξάρτητο φορέα στα κράτη-μέλη. Τώρα, έχουμε, μπορούμε ευθέως να πούμε ότι δεν θα πρέπει ο φορέας πιστοποίησης να υπάγεται ευθέως στον ε, διευθυντή του οργανισμού πληρωμών. Ναι βεβαίως, αλλά από τη στιγμή που ένας τέτοιος οργανισμός βρίσκεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, μιας εθνικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πει τίποτα από αυτού. Η νέα ΚΑΠ θα είναι πιο απλή ή πιο περίπλοκη. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία απλοποίησης των διαδικασιών. Στον τομέα της ανάπτυξης της υπέρθρου σας τα ανέφερα μερικά από αυτά τρόπο με τον οποίο ορίζονται τα μέτρα, τα που τώρα είναι ε, πιο καλά ορισμένα, γιατί γνωρίζετε πολλές φορές η πολυπλοκότητα προερχόταν από ασαφείς ορισμούς. Τώρα οι ορισμοί του δεύτερου πυλώνα είναι πιο σαφείς και αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, έχουμε πλέον στοιχεία που δεν είχαμε στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα την καθυστέρηση ε, των πληρωμών. Αλλά και αυτή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ελέγξιμο. Οφείλουμε να λογοδοτούμε για τα χρήματα που δίνονται μέσω των άμεσων πληρωμών στους αγρότες. Και αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι οι αγρότες θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση αυτών των χρημάτων. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε οι απαιτήσει οι οποίε επιβάλλουμε στου αγρότε θα είναι αρκετά απλέ, έτσι ώστε να μπορούμε και εμεί να ελέγξουμε κατά πόσον τη στήρισαν. Για παράδειγμα, στο ζήτημα τη επιλεξιμότητα, όχι μόνο για τι χορτοδηλευαστικέ εκτάσει τη μόνιμε, αλλά ιδιαίτερα για αυτέ, τώρα πια ο ορισμό αυτών των εκτάσεων είναι πολύ πιο απλό, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούμε να ε, διεξάγουμε ελέγχου απλούστερου και πιο αποτελεσματικού. Αυτό μπορώ να σας πω. Τώρα, αν το επιθυμείτε, μπορώ να σας προετοιμάσω ένα έγγραφο που να καταγράφει ε, συγκεκριμένα ποιες είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα στοιχεία απλοποίησης κατά πυλώνα. Τώρα, εσείς ε, ε, ε θέτεται συνέχεια θέματα για την Ελλάδα και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των χρηματών στην Ελλάδα και το σύστημα οριοθέτηση των γεών. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, αλλά έρχομαι στη Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει ε, καταβάλει μια σημαντική ε, δημοσιονομική διόρθωση και επίσης ε, έφτιαξε από την αρχή τη βάση δεδομένων το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και διαπιστώνουμε τώρα ότι το σύστημα για τον πρώτο πυλώνα λειτουργεί. Για το δεύτερο πυλώνα έχουν ήδη διαπιστωθεί τα προβλήματα σε διάφορα μέτρα, η ποιότητα των ελέγχων σε διάφορα μέτρα και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία ε, διατύπωση, επαναδιατύπωσης μάλλον των κριτηρίων επιλεξιμότητας και έχει υπάρξει αναστολή πληρωμών μέχρι να γίνει ο έλεγχος επί 2-3 μέτρων που μας έχουν προβληματίσει. Χωρίς αμφιβολία θα υπάρξει επιβολή επίσης και δημοσιονομική διόρθωση στον δεύτερο πυλώνα. Αλλά όπως σας είπα για τον πρώτο πυλώνα, μετά τους ελέγχους που διεξάγαμε, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το σύστημα λειτουργεί και ότι τα προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί εξαιτία τη ε, μη επαρκούς ποιότητας των ελέγχων έχουν πλέον διορθωθεί. Λίγα ήταν εκείνα της κελιός για τον πρώτο πυλώνα γιατί δεν επρόκειτο για συστημικά προβλήματα, αυτά διορθώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, στη, στη, στο δεύτερο πυλώνα, στη Ρουμανία, εξετάζουμε ενδελεχώς την κατάσταση. Okay, merci Σας ευχαριστώ. Α, πρέπει να κοιτάξουμε και την ώρα. Ήθελα όμως να ρωτήσω αν το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάποιες ερωτήσεις. Ε, κύριε Κούμπικ, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος, κυρίες και κύριοι. Τρεις εξηγήσεις ε, και ένα συμπέρασμα για την μεθοδολογία μας. Δεν ε, έχει αλλάξει μεθοδολογία σε σχέση με το κεφάλαιο 3 και 4 της ετήσιας έκθεσης. Οπότε ε, οι εκθέσεις του 11 και του 12 είναι συγκρίσιμες. Όσον αφορά την δειγματοληψία μας, ε, το βλέπετε στην υποσημείωση 21 του κεφαλαίου 3. Το ελεγκτικό συνέδριο υπολογίζει το ποσοστό σφάλματος με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και έχουμε 95% εμπιστοσύνη πώς βρισκόμαστε μεταξύ του ανώτερου και του κατώτατου ποσοστού. Αυτά στο παράδειγμα 1 του κεφαλαίου 1. Όσον αφορά το ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ συνεχίζει να έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό σφάλματος. Μπορεί να δει τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ μαζί με, ε, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ένα πράγμα όμω το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι πως κανένα σύστημα δεν είναι δεδομένο για πάντα. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να αποφύγουμε, όπως είπα, τον επηρεαστεί το σύστημα από ανακριβείς βάσεις δεδομένων. Και τέλος, συμπρασματικά θα ήθελα να πω πως αναμένω τις περαιτέρω βελτιώσεις στην διαχείριση της γεωργίας, ειδικά με την εφαρμογή των συστάσεων του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρία δεν θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα μόνο να πω πως για την ανάπτυξη της υπαίθρου το το είναι πάνω από το 2% του επέδου σημαντικότητας. Και τέλος, ε, μεγάλο τμήμα των απαντήσεων του Επιτρόπου βεβαίως στις αδυναμίες που σημειώσαμε είναι πως το σχέδιο δράσης ε, και η περισσότερη προσοχή που θα δοθεί στις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις θα βοηθήσουν στη μείωση του ποστού σφάλματος. Το ελεγκτικό συνέδριο θα παρακολουθήσει την κατάσταση, σας διαβεβαιώ πάρα πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Πίπερ, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή... Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω για την ε, συζήτηση αυτή όλους. Και οπωσδήποτε θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης.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 to not. Θα uh, προσθέσω να είμαι στο δυνατόν πιο σύντομος. Γκέρχαρτ Σμιτ λέγομαι από το Οικολογικό Ινστιτούτο. Μας έδωσε εντολή η Επιτροπή του Προϋπολογισμού να προετοιμάσουμε μία μελέτη Οπότε με στόχο να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, κλεισίματος των εργοστασίων στην Ευρώπη. Το δεύτερο ήταν να περιγράψουμε και να συγκρίνουμε τις διαδικασίες στη Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία που ε, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις συγκρίνουμε με άλλες βέλτιστες πρακτικές και τέλος και είναι το βασικό. Ε, να κάνουμε συστάσεις για βελτίωση της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για τις βέλτιστες πρακτικές. Είχαμε το εξής αποτέλεσμα. Έχουμε 88 αντιδραστήρες ε, που είναι σε διαδικασία πάυσης ε, λειτουργίας διαφόρων τύπων και μεγεθών. Περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στη Γαλλία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και η επιχειρησιακή τους ε, ηλικία επίσης κυμαίνεται από λίγα χρόνια μέχρι πάνω από 40 χρόνια σε κάποιες ε, περιπτώσεις και από τους 88 αντιδραστήρες μόνο 8 έχουν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η πάυση λειτουργίας τους. Οπότε το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι πως ε, δεν έχουν ε, οριστικοποιηθεί τα έργα αυτά, οπότε αν αναζητήσετε αποτελέσματα για το κόστος και τέτοια πράγματα, κυρίως μιλάμε για υποθέσει. υποθέσεις, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σοβαρά. Τρία παραδείγματα εξετάσαμε πιο προσεκτικά της Electricité de France που αυτή τη στιγμή βγάζει εκτός εννέα αντιδραστήρες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, αλλά με κύριο μετοχό το κράτος. Οι δε νέα αντιδραστήρες ε, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία από το 2002, πριν από 11 χρόνια. Μετά είχαμε την Ενεργή Ιβέρ και Νόρντ, μια εταιρεία που ανήκει στο Ομοσπονδιακό Δημόσιο της Γερμανίας. Ε, έξι αντιδραστήρες ε, είναι υπό απόσυρση τύπου συγκρίσιμου με τις Βουλγαρίας και τις Σλοβακίας. Και μετά κοιτάξαμε και την Σέλαφιλντ ΑΕ ε, μεγάλη εταιρεία βρετανική υπό τον έλεγχο της ε, Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας η οποία ελέγχει πολλές εγκαταστάσεις. Οι βέλτιστες πράκτικες που βρήκαμε ήταν οι εξής, πως πρέπει να υπάρξει πλήρης αναδιοργάνωση οργανισμών οι οποίοι θα έχουν την καταλληλότερη μορφή για απόσυρση των εγκαταστάσεων. Το να κάνουν οι ίδιοι την λειτουργία και την απόσυρση δεν οδηγεί σε βελτιστή λειτουργία. Αυτό κατέστη σαφές στην ΕΔΕΦ της Γαλλίας και στην ΕΒΕΝ της Γερμανίας Οπότε η οργανωτική δομή έπρεπε να προσαρμοστεί πλήρως στην απόσυρση αντί να ε, είναι η ίδια με την δομή της κανονικής λειτουργίας. Το δεύτερο συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως έπρεπε να ελέγχουμε στενά τις ε, στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης που θα εξετάζει λεπτομερώς όπως είπα τις αποφάσεις αυτές ε, στην περίπτωση αυτή αυτός ο φορέας ήταν το Υπουργείο Οικονομικών ε, της Γερμανίας στην EDF ε, ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Το επόμενο το οποίο είδαμε είναι πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα πλήρες εργαλείο διαχείρισης έργου και κάποιες αρχές διαχείρισης έργου κατά τη διάρκεια της απόσυρσης. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό βέβαια από τη φάση κανονικής λειτουργίας όπου τα πράγματα πάνε σύμφωνα με το εχειρίδιο ε, που ε, κάθε ενέργεια περιγράφεται σε αυτό και απλά ακολουθεί κανείς αυτές τις οδηγίες πάρα πολύ ε, στενά. Στη, για τη διαδικασία της απόσυρσης δεν υπάρχει εγχειρίδιο, δεν υπάρχει κάτι το τυποποιημένο οπότε με το να έχουμε όπως είπα διαχείριση του έργου αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη και στη Γαλλία και στη Γερμανία και τη διαχείριση αυτή την περιγράφουμε λεπτομερώς στη μελέτη. Το τέταρτο που πρέπει να αναφέρουμε είναι πως η απόσυρση πρέπει να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει το εργατικό δυναμικό το οποίο λειτουργούσε τον αντιδραστήρα μικρή πρότινος να χρησιμοποιήσει την γνώση τους τη γνώση που έχουν για τις εγκαταστάσεις αλλά θα πρέπει βεβαίως να επανεκπαιδευτούν για την δουλειά της απόσυρσης. Μετά συγκρίναμε τα ζητήματα αυτά που ανέφερα με την κατάσταση στη Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία. Ελπίζω να είναι έγχρωμο το διάγραμμα αυτό, ωραία ναι. Βλέπετε λοιπόν από το άριστα, το οποίο είναι 5, ειδικά το εθνικό πλαίσιο, ε, την οργάνωση της διαχείρισης ε, και τη διαχείριση έργου και κινδύνου πλην Σλοβακίας, ε, βλέπετε πως έχουμε αρκετό περιθώριο βελτιώσεων. Ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες δηλαδή ρυθμιστική προσέγγιση, εκτίμηση του κόστους και το εργατικό δυναμικό είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να έχει εργατικό δυναμικό ε, υπάρχει ακόμα κάποιο περιθώριο. Οπότε, τι βρήκαμε στη σύγκριση αυτή, πως ε, το εθνικό πλαίσιο μπορεί να βελτιωθεί σε Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία. Και κυρίως τα ζητήματα βεβαίως εντοπίζονται σε Βουλγαρία και Λιθουανία. Οι φορείς οι εθνικοί οποίοι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για την απόσταση δεν έχουν την ε, ιδανική οργάνωση για να αναλάβουν το καθήκον αυτό και επίσης η διαχείριση όπως είπα μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ. Καταλήξαμε σε 8 συστάσεις τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στη μελέτη ειδικά τα σημεία 8 για την σαφή κατανομή των ευθυνών για ε, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, αυτή είναι η πρότασή μας για την ε, αναδιάρθρωση της ε, διοίκησης της Εθνικής Υπηρεσίας Απόσυρσης και Βλέπετε εδώ πέρα πάει σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας ποιος πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις σε ποιο επίπεδο. Το επίπεδο αποφάσεων είναι τόσο στρατηγικό και το επιχειρησιακό και οι επιχειρησιακές αποφάσεις πρέπει σαφώς να λαμβάνονται από το διαχειριστικό επίπεδο του οργανισμού ενώ οι στρατηγικές αποφάσεις ε, από την εθνική διοίκηση και την κοινότητα. Αυτή είναι η βασική μας πρόταση για την αναδιάρθρωση της ε, διαδικασίας απόσυρσης και είμαι σίγουρος πως με αυτή την αναδιάρθρωση μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σμιτ για την παρουσίαση των ουσιαστικών αποτελεσμάτων της μελέτης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Το, με συγχωρείτε στον εισηγητή πρώτα. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Εσείς και οι συνεργάτες σας ε, ταρακουνήσατε τα λιμνάζοντα ύδατα. Η νομοδότηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ε, κάτι που έχουμε λάβει και βεβαίως έχουμε και την δική σας την αντίδραση που ξεκαθάρισε κάποια πράγματα προφανώς αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα γιατί όπου ανακοινείται η κατάσταση κάτι που όπου ταράζουν τα ύδατα κάτι δεν πήγαινε καλά στο παρελθόν. Προσδήποτε λοιπόν θα πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τώρα, σε λίγο θα ξεκινήσουν οι δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Πάλι θα έχουμε 816 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δουλειά. Το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα λεφτά είναι ένα θέμα στο οποίο θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να έχουμε κάποιο λόγο. Ως ε, Επιτροπή Ελέγχου του Περιπολογισμού έχουμε ταξιδέψει και στα τρία αυτά μέρη, εγώ δυστυχώς μόνο στα δύο, αλλά οι συνάδελφοι ε, έχουν πάει σε όλα, οπότε έχουμε μία κάπως συνολική εικόνα Έχω όντως μια ουσιαστική ερώτηση. Μιλήσατε για τις βέλτιστες πρακτικές ε, ε, στις οποίες δεν συμπεριλάβατε τη Γαλλία. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πως βγάλατε ένα κομμάτι από τις βέλτιστες πρακτικές χωρίς μικρόφωνο ο Σμιτ. Κάναμε την περιγραφή, ή μάλλον δεν κάναμε την περιγραφή τριών ε, στοιχείων τα οποία αξιολογούμε στην παρούσα παρουσίαση. Αλλά το κάνουμε αυτό στη μελέτη, λεπτομερέστερα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση την οποία μόλις σας έκανα και η οποία υποχρεωτικά έπρεπε να είναι σύντομη και στο σύνολο της μελέτης και τις αναφορές στη μελέτη. Εμείς εξετάζουμε λεπτομερώς και την γαλλική περίπτωση και την γερμανική περίπτωση και κάνουμε μια κατανομή θα έλεγα στον χώρο περίπου ισότιμη. Μάλιστα. Είμαστε εδώ πέρα την ε, σύνοψη είπατε πως ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παρουσίαζε ε, πάρα πολλά πλεονεκτήματα ως παράδειγμα προς Ποια είναι η διαφορά εκεί πέρα. Μετά. για να επανέλθω στο θέμα της ασάφειας της ευθύνης. Γιατί αναφέρατε κάποια παραδείγματα. Εμείς είχαμε την εντύπωση πως ε, από τα τρία έργα που εξετάσατε η ευθύνη και άρα η επιτόπια διαχείριση ε, είναι καλύτερη στην ε, Σλοβακία, δηλαδή η αρχή εκεί πέρα, η Γιάρης, όπως λέγεται, για την απόσυρση των πυρηνικών αυτών εργαστοσύνων είναι μια κρατική επιχείρηση και βεβαίως εντάξει, υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι το ότι είναι κεντρική η διοίκηση και ο κίνδυνος βεβαίως θα μπορούσε να είναι πως ε, ως ε, κρατική ε, εταιρεία στην ανάγκη δεν θα είναι ανεξάρτητη και όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε όταν έχουμε διαγωνισμούς δεν είναι σαφές ε, το τι αγοράζουμε με τα λεφτά μας αν θέλετε. Δηλαδή δεν ε, ακολουθούν αυστηρά θα έλεγα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ε, οικονομίας όπως θα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς το βλέπετε εσείς ε, τα υπέρ και τα κατά δηλαδή μιας έτσι τόσο συγκεντρωτικής αρχής και ε, προτάσεις για αξιολόγηση και μετά έχουμε νομική βάση για κάτι τέτοιο ή τι θα έπρεπε να κάνει το κοινοβούλιο να απαιτήσει από την Κομισιόν ως μέσα για να εφαρμοστεί μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε αμέσως, παρακαλώ. Ναι, ναι, πριν ξεχάσω. That is very relevant. Νομίζω ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σχέση το πώς θα το εάν θα έχει δομή ιδιωτική εταιρεία ή δημόσιου φορέα αυτός ο φορέας και στην περίπτωση της CDF και στην περίπτωση της CWN ήταν διαφορετική η δομή αλλά εξίσου αποτελεσματική. Στη Γερμανία το Υπουργείο Οικονομικών ελάμβανε τις στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας. και αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μη αποτελεσματική η δομή απόσυρσης. Ούτε οδήγησε σε υπερτιμολογήσεις. Δεν συνέβη αυτό στη Γερμανία. Και δεν συνέβη παρά το γεγονό ότι πρόκειται για μια δημόσια ε, επιχείρηση Η EDF από την άλλη, ιδιωτική εταιρεία, ούτε εκείνη υπήρξαν αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται η απόσυρση των πυρηνικών αντιδραστήριων με ε, δημόσιους φορείς αντί για ιδιωτικές εταιρείες. Δεν σημαίνει αυτομάτως ή αμέσως ότι είναι αυτές οι ε, δομές αποτελεσματικότερες. Το θέμα είναι η δομή τους. Εάν σε αυτή την εταιρεία αποδοθούν σημαντικές αρμοδιότητες και, θα έχει, και να, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις, τότε θα λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις. Εάν όμως δεν συμβεί αυτό, ο φορέας που ασκεί τον έλεγχο, συνήθως το Υπουργείο, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του εξίσου. Και να ασκεί μικροδιαχείριση όσον αφορά αυτό το φορέα. Ως κανόνα λοιπόν διαπιστώσαμε και στην EWM και στην EDF ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθεί όσο το δυνατό περισσότερο το εργατικό δυναμικό του ιδίου του φορέα της απόσυρσης. Με άλλα λόγια, να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο οι εξωτερικοί συνεργάτες. Γιατί είναι πιο αποτελεσματικό να ενισχυθούν τα προσόντα του εργατικού δυναμικού του ίδιου του φορέα και να αναλάβει το ίδιο το προσωπικό της διάφορες εργασίες, παρά να ασχολείται ο υποπτεύων φορέας με τις λεπτομέρειες ε, της διοίκησης και, και, του έργου αυτού του φορέα. Καλύτερα ο υποπτεύων φορέας να ασχολείται με τους γενικούς κανόνες, για παράδειγμα, για τις δημόσιες συμβάσεις, για την προμήθειες κτλ. Και τα δύο παραδείγματα, το γαλλικό και το γερμανικό, ε, είναι ε, θετικά. Σε αντίθεση με αυτά τα δύο παραδείγματα μπορούμε να δούμε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ανατέθηκε σε εξωτερική εταιρεία η ε, απόσυρση. Μόνο, υπάρχει μόνο ένας εμποπτεύων φορέας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες. που έχουν, περιορισμένη ευθύνη για τυχόν λαθασμένες αποφάσεις ή πράξεις τους. Και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα. concerns uh, όσον αφορά τα έργα τα οποία βρίσκονται σε κοινή διαχείριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, με τους αρμόδιους φορείς τους. Πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Έτσι θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα γιατί ενισχύεται ο ρόλος του, ε, δημόσιου, του φορέα στο κράτος μέλος να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η Σλοβακική αρχή μας δίνει ένα καλό παράδειγμα γιατί πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση τα περισσότερα από τα έργα που θα υλοποιηθούν στη Σλοβακία βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σλοβακίας. Η Γιάβης λοιπόν είναι μια από τις ε, πιο αποτελεσματικές από τους πιο αποτελεσματικούς φορείς απόσυρσης που έχουμε δει. Ja, vielen Dank. Jetzt... Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φάζακας από το Ελληνικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση και μας δώσατε δυνατότητα να τοποθετηθούμε ε, για αυτή τη μελέτη και γενικά για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εξ μου και εξ ονοματός του Ελεκτικού Συνεδρίου εσάς ε, και τον κύριο Γιάννη Σκάιερ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για το ότι ζητήσατε αυτή την ε, μελέτη του Οικολογικού Ινστιτούτου και την ε, βάλατε σήμερα στην μερίσια διάταξη. μελέτη αυτή δεν έκανε μόνο κάποιες σημαντικές διαπιστώσεις και συστάσεις ε, όσον αφορά την απόσυρση των πυρνικών εργοστασίων σε Βουλγαρία, Λιθουανία και αλλού, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήδη ως εγχειρίδιο. Ήδη αναφέρατε πως 88 αντιδραστήρες βρίσκονται σε διαδικασία κλεισίματος και θα ακολουθήσουν εκατοντάδες. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει κάποια αρμοδιότητα σχετική στο μέλλον. Αλλά γενικά θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και την αναγνώρισή μας για το ότι η Επιτροπή σας ανέλαβε την πρωτοβουλία να δει αυτό το σημαντικό ζήτημα. Για να δούμε τα γεγονότα των τελευταίων ετών, διαπιστώνουμε πως η Επιτροπή Ελέγχου του Υπερπολογισμού είχε θέσει πριν από πέντε χρόνια το ερώτημα του εάν γίνονται όλα σωστά στην, στις αποσύσεις, εάν τα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής ε, ευρωπαϊκών εισφορών χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για να λάβουμε μία απάντηση. Ζητήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει μία σχετική μελέτη και έκθεση. Το ελεγκτικό συνέδριο δέχτηκε ευχαρίστως και μετά από λεπτομερή εξέταση εγκρίναμε μία ειδική έκθεση το 2011. Η έκθεση αυτή 16-2012 ήδη εγκρίθηκε από την Επιτροπή σας οπότε τώρα δεν θεωρώ πως είναι η στιγμή να αναφέρουμε τα ευρήματα και τις συστάσεις μας. Αρκεί να πούμε αυτό το οποίο αναφέρεται στην έκθεση πως διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα μπορούσε ε, βεβαίως ε, να πούμε πως ε, πρέπει να υιοθετήσει τις συστάσεις μας η Κομισιόν και βεβαίως ε, η Επιτροπή σας, ε, όπως είπαμε, δεν κόπον είναι για να πάει επί τόπου και να διαπιστώσει στην πράξη πώς εφαρμόζονται οι συστάσεις μας. Τώρα, μετά από πέντε χρόνια, διαπιστώνουμε και μπορούμε να ισχυριστούμε πως τουλάχιστον ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Πρώτον, διαπιστώνουμε με χαρά και ικανοποίηση πως με, λόγω της ευρωπαϊκής συνεισφοράς ήδη έχουν κλείσει πλέον αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια και η διαδικασία αυτή δεν αναστρέφεται. Πρέπει να τονίσουμε αυτό γιατί δεν ήταν καθόλου σίγουρο. Οπότε ο βασικός στόχος, η πυρηνική ασφάλεια, έχει επιτευχθεί. Επιπλέον ξέρουμε και αυτό φαίνεται και στην μελέτη το ποια σημαντικά πράγματα έχουμε να κάνουμε, ποιο κόστος έχουν, γνωρίζουμε πως παρά το ότι ε, στην επόμενη περίοδο προβλέπονται 860 εκατομμύρια θα έχουμε μεγάλα κενά ταυτόχρονα αναδείχτηκαν σημαντικά οργανωτικά προβλήματα που είναι τόσο σημαντικά ώστε επηρεάζουν την έγκαιρη ε, ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου κόστους. Οπότε απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Αναφερθήκατε και κάνατε 8 σημαντικές προτάσεις ε, βελτιώσεων και βεβαίως πρώτον δεν είναι δουλειά του Ελεκτικού συνεδρίου να αξιολογήσει αυτές τις προτάσεις όταν εφαρμοστούν θα ε, εκφράσουμε την απόψή μας για την εφαρμογή αλλά τέλος ε, θα θέλαμε να τονίσουμε σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γιέντς Γκάιερ πως ανεξαρτήτως του ποια οργανωτική δομή επιλεγεί και εφαρμοστεί η τελική ευθύνη στην εφαρμογή και στην χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι της Κομισιόν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η Κομισιόν είναι ο ελεγχόμενος, η Κομισιόν είναι ο συνομιλητής της Επιτροπής σας και εδώ πέρα πρέπει να ακούσει αυτά τα οποία λέτε και να τα εφαρμόσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Σε ποιον να δώσω λόγο για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα Είμαι η Τάρχης στη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με το θέμα. Θεωρούμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δυστυχώς οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Λουξεμβούργου που έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, α, έφτασαν δεν μπορούσαν να έλθουν. Εν περιπτώσει δεν ξέρω, έχει δημιουργηθεί μια παρανόηση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα τις σημειώσουμε και θα σας απαντήσουμε. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορέσαμε να είμαστε σε θέση να πάρουμε μέρος στη συζήτηση. Ε, μου είπαν ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας δεν έχει ακόμα φτάσει, αλλά βλέπω ότι είναι εδώ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι είμαι εδώ. Θα συνεχίσω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Η έκθεση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση της το θέμα της εφαρμογής και χρήσης μάλλον των πιστώσεων είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας και είναι υποχρέωση για τις υπηρεσίες μας να συνεργαστούμε σωστά προς την κατεύθυνση αυτή. Μετά από την πρώτη ανάλυση που κάναμε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιες σημαντικές επιφυλάξεις σε κάποια τεχνικά θέματα. είμαστε σαν υπηρεσία σε θέση να κρίνουμε τεχνικά κάποιες πλευρές και θα σταθώ σε αυτές. Πρώτον, το θέμα της συνολικής παρουσίασης που ε, ελείπει για μας θα πρέπει να περιγραφεί θα έλεγα καλύτερα το πλαίσιο το πολιτικό πλαίσιο και το οργανωτικό για κάθε χώρα και σε επίπεδο κυβερνητικό και σε επίπεδο διοικητικό ε, για τις πυρηνικές μονάδες. Ε, επίσης το θέμα των αλλαγών με το χρόνο. Υπήρχε μια πολύ σημαντική έκθεση του 11 του ελεγκτικού συνεδρίου που έδωσε συγκεκριμένες συστάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν γρήγορα και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να δώσουμε μια ε, εικόνα του πού βρίσκεται η κατάσταση, αλλά να μετρήσουμε και τις συνέπειες της απόφασης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Ήδη εμείς βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές. Δύο επιπλέον παρατηρήσεις τις οποίες επιλέγω ανάμεσα σε άλλες. Επιλέγουμε χώρες όπου υπάρχουν ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό παροπλισμό, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές διαφορές ε, για τις επίπεδο πληροφοριών. Βλέπουμε ότι για τη Γερμανία έχουμε πολλές πληροφορίες ενώ για άλλες χώρες όχι. Είναι δύσκολο να κρίνει κανείς λοιπόν αν μπορεί να προχωρήσει σε ανάλυση με ομοιογενείς πληροφορίες. Η Γαλλία δεν έχει ολοκληρώσει τον αφοπλισμό και στο Ηνωμένο Βασίλειο το Calder Hall είναι μια μικρή πυρηνική μονάδα ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας ευρύτερης πυρηνικής μονάδας του Σέλαφιλντ. Υπάρχουν στην έκθεση κάποιες αρνητικές κρίσεις σε σχέση με τη μείωση του μεγέθους των υλικών και του εξοπλισμού που έχει αυτή τη στιγμή αποσυρθεί. Τεχνικά ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν στέκει γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το ότι ε, πριν προχωρήσουμε ε, στις διαδικασίες αυτές είχαμε κάνει και είχε γίνει και μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαχειριστική ομάδα τμήμα του συνόλου της επιχείρησης αφοπλισμού μιας μονάδας ε, δεν έχει γίνει κάτι το κατανοητό. Και νομίζω ότι κάποια από τα συμπεράσματα λοιπόν δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της EBRD, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, ε, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Συμφωνώ με την εισαγωγή την οποία έκανε ε, ο συνάδελφος. δεν είναι σωστό το να αναμειγνύει κανείς τα θέματα της λειτουργίας μιας πυρηνικής ομάδας με το θέμα του αφοπλισμού, του παροπλισμού συγγνώμη, της συγκεκριμένης μονάδας. Υπάρχει, υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά στην διαδικασία παροπλισμού της μονάδας. Φυσικά και πρέπει να εμπλέξουμε το προσωπικό το οποίο συμμετέχει ε, στην ε, λειτουργία της μονάδας. Με αυτό συμφωνούμε 100% όμως το βασικό σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω για την έκθεση είναι ε, τα δεδομένα στα οποία βασίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη και δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε σοβαρά τις συστάσεις. Να υπογραμμίσω κάποια από αυτές ε, τις ελλείψεις, να ξεκινήσω τις, από την παρουσίαση η οποία περνάει από τα βασικά στοιχεία ε, στα benchmark και βλέπετε κάποια γραφικά τα οποία είναι πιστικά αλλά είναι αστήρικτα από την άλλη. και για κάποιες από τις χώρες ε, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πραγματικά υβριστικά. Τι θέλω να πω. δεν κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στη διαχείριση της μονάδας και στη διαδικασία παροπλισμού της, ομάδας, της μονάδας. Είναι κάτι ο παροπλισμός που πρέπει να γίνει από συγκεκριμένους οργανισμούς ελεγχόμενους από τις κυβερνήσεις. Δεν κάνουν τη διάκριση λοιπόν ανάμεσα στις ε, επιχειρήσεις αυτές και στις κυβερνήσεις οι οποίες καλούνται επίσης να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο χρήμα. σχετικά με τη διαχείριση, την διακυβέρνηση της διαδικασίας παροπλισμού εδώ τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί η έκθεση είναι λανθασμένα. Να σας δώσω κάποια απλά παραδείγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγιναν αυτά τα λάθη. Μία χώρα η οποία παίρνει αυτή τη στιγμή χρήματα για τον παροπλισμό ε, λέει η έκθεση ότι είναι απλώς παρατηρητής. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Ε, κάθε κυβέρνηση έχει ε, πλήρεις αρμοδιότητες και δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Λέει ότι η τράπεζα προετοιμάζει ε, η τράπεζα για την ανάπτυξη και την... The report says the PMU consultant has a contract with the EBRD. Not true. Λέει λοιπόν ότι η τράπεζα είναι αυτή τα οποία προετοιμάζει, αυτό δεν είναι αλήθεια γίνονται προγράμματα και αφού η διαχειριστική εταιρεία έχει κάνει τις προτάσεις της αποφασίζεται για το τι περαιτέρω προσπάθεια απαιτείται και τι μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη απαιτείται με βάση τις προσφορές. Και τέλος και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Η έκθεση λέει ότι το PMU είναι εκτός της διαχειριστικής μονάδας. Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι τμήμα της διαχειριστικής μονάδας. Δηλαδή το σχέδιο της παρουσίασης είναι λανθασμένο, είναι αστήρικτο. Όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικέ συνθήκες οι οποίες επικρατούν στις τρεις χώρες και τη διαδικασία παροπλισμού που κρατάει κάποια χρονική περίοδο. Υπάρχουν διαδικασίες κλεισίματος, υπάρχουν ε, τα προβλήματα της αντίδρασης σε αυτό, η σοβιετική κληρονομιά, η συνέχιση σε ορισμένες περιπτώσεις της λειτουργίας μονάδων, Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη και επηρεάζουν αρνητικά ε, και τα benchmarks τα οποία περιγράφονται εδώ με άδικο και ατελή τρόπο. Και όπως είπε προηγουμένως και ο μιλητής, δεν λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις από τότε που έγινε, δημοσιεύθηκε η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρόκειται για ευρήματα τα οποία κυκλοφόρησαν εδώ και τρία χρόνια και θα έλεγα οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το παράδειγμα της μονάδας τήξης πλάσματος στη Βουλγαρία που η έκθεση θεωρεί ότι είναι παράδειγμα κακής διαχείρισης και χρησιμοποίηση μη τεκμηριωμένων τεχνολογιών. Αυτό είναι λάθος. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία ισχύει, κάποιοι έχουν διαφορετικές απόψεις, αυτό είναι φυσιολογικό στα πλαίσια της βιομηχανίας. Ένα αντίστοιχο κέντρο λειτουργεί πολύ καλά στην Ελβετία και το χρησιμοποιούν επιχειρήσεις ε, ε, πολύ σημαντικές και σεβαστές σε διάφορες χώρες μέλη. Τα θέματα των διαγωνισμών επίσης ε, και των προμηθειών και αυτά παρουσιάζονται με εντελώς λανθασμένο τρόπο. Οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε ιδιαίτερα στα πλαίσια της δικής μου τράπεζας γίνονται με βασικό στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών. Οι τελευταίοι έλεγχοι που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασαν και τις συμβάσεις που φτάνουν τα 885 εκατομμύρια ευρώ και δεν βρήκαν τίποτα το αρνητικό. Αυτά σχετικά με την προστασία του δημόσιου χρήματος. Δεν βρέθηκε κανένα πρόβλημα στα πλαίσια της λειτουργίας αυτού του προγράμματος. Συμπερασματικά, η έκθεση που παρουσιάστηκε εδώ δεν δίνει καμία σωστή ανάλυση της επίδοσης των προγραμμάτων, βασίζεται σε τεκμήρια λανθασμένα, σε απλούς ισχυρισμούς και ως εκ τούτου είναι λογικό τα, συμπεράσματα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει να είναι εντελώς μοιραία λανθασμένα. Ευχαριστώ. Τώρα Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Η κυρία Γκρέσλε βεβαίω έχει ζητήσει το λόγο. Ε, είχα υπομονή γιατί είναι σημαντική η συζήτηση. Καλό θα ήταν το Ινστιτούτο να τοποθετηθεί για όλα αυτά. Θεωρώ πως για εμάς εδώ πέρα στη Λιθουανία το... η Λιδία Λίθος είναι η Γναλίνα ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορέσουμε να κρίνουμε όταν ολοκληρωθεί βέβαια η διαδικασία. Τώρα είμαστε κάπου στη μέση. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω πως ε, δεν είχε εκεί πέρα οργανωθεί η διαδικασία της ε, απόσυρσης ε, με κοινή διαχείριση έτσι όπως έχουμε στα διαρθρωτικά ταμεία. Γι' αυτό κατά την άποψή μας και σωστό είναι αυτό. Κάποια συμπεράσματα τα βρίσκω πάρα πολύ γενικά. Είναι, δηλαδή μοιάζει σαν να τα έχετε αντιγράψει από κανένα εγχειρίδιο οικονομικών. Ναι, εντάξει, πράγματι. Καλό είναι να υπάρχει σαφής ε, διοικητική δομή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αλλά όταν έχουμε πολλούς ε, φορείς... Ε, και περιπλοκές δομές και επιπλέον ε, ένα φορέ ελέγχου ξεχωριστό όπως είναι η Κομισιόν. Ε, έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω πως λειτουργούν αρκετά καλά δεδομένα των ε, συνθήκων. Εγώ έχω επισκεφθεί και τα τρία εργοστάσια. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την επαγγελματική επάρκεια των εργαζομένων. Αυτό το οποίο αμφισβητώ είναι η σοβαρότητα του κράτους μέλους ε, να τα κλείσουν και να χρησιμοποιήσουν τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια που διαθέτουν. Γιατί, τι λένε, όσο περιμένουμε τόσο περισσότερα λεφτά έρχονται. Έτσι, οπότε... Τελικά δεν θα έχουμε ποτέ ένα οριστικό κλείσιμο. Τέλος αν δεν έχω διαβάσει ακόμα ολόκληρη τη μελέτη, θα το κάνω. Αλλά Είμαστε στη μέση της διαδικασίας, οπότε αντιλαμβάνουμε τα προβλήματα τα οποία λέτε. Η μελέτη ταυτόχρονα είναι και πολύ νωρίς και πολύ αργά, ε, ε, η χρονική στιγμή στην οποία έρχεται. Έχει πολλές γενικότητες, γι' αυτό δεν μπορώ τώρα να πω πως ναι εντάξει μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την διαδικασία. Για εμένα είναι σημαντικό να δούμε το θέμα της ευθύνης. Γιατί κοιτάξτε, άμα πάνε στραβά τα πράγματα στην ε, Ιγναλίνα, ξέρετε θα πούνε, «Ε, το κοινοβούλιο τότε τι έκανε. Δεν παρατηρούσε τίποτα. Για μένα λοιπόν πραγματικά η Ιγναλίνα είναι το, το βασικό ζήτημα. Το Κοσλοντούι λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά στην ημερήσια διάταξη. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω διαβάσει ακόμα την απάντηση της ε, βουλγαρικής κυβέρνησης. Και νομίζω αυτά είναι μεγάλες ε, επιτυχίες. Ε. Δεν ξέρω πραγματικά ανησυχώ και για τον επαγγελματισμό και για την θέληση. αν υπάρχει όντως θέληση να κλείσει αυτός ο σταθμός. Και δεν ξέρω πραγματικά όντω αν υπάρχει κάποια προσθέμενη αξία στη μελέτη αυτή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ να είστε και λίγο σύντομοι. Ο κύριος Κάλβιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι ακούσαμε <clears throat> από την Επιτροπή και από την Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης μου δίνει τη δυνατότητα να περιορίσω και τις παρατηρήσεις μου στο ελάχιστο. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι χρήσιμη γιατί θέτει κάποια ερωτήματα. Τουλάχιστον ε, έχουμε ένα ζήτημα να συζητήσουμε εδώ. Τα στοιχεία όμως που αναφέρονται κάποια από αυτά δεν είναι σωστά, κάποια, παλιά, κάποια είναι παπαλαιωμένα. Αναφέρεστε για παράδειγμα σε προ παρασκευαστικές εκθέσεις του 2008 ενώ η τελική έκθεση δημοσιεύτηκε το 2011 και δεν ελήφθη υπόψη. Τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα αλλά εγώ θα σταθώ στα σημεία που, θεωρώ, σημαντικά για το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Πρώτα απ' όλα είναι το ζήτημα του κατά πόσο υφίσταται μια σωστή δομή για να διαχειριστεί τη διαδικασία παροπλισμού. Δεν γνωρίζουν την κατάσταση σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, όμως νομίζω ότι μία από τις κριτικές που εκφράζεται εδώ έχει ήδη, ε, είναι ήδη παροχημένη γιατί έχουν ξεχωριστεί οι δομές, ίσως ίσχυε πριν 3-4-5 χρόνια, αλλά δεν ισχύει πλέον αυτό. Υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο σύστημα διοίκησης, μια ξεκάθαρο σύστημα λογοδοσίας και μια ξεκάθαρη δομή Είχαμε πολλές συζητήσεις σε θεσμικό επίπεδο με πολλά γραφήματα κτλ. Το PMU είναι πλέον μέρος της μονάδας διαχείρισης και αυτό έχει αλλάξει την κατάσταση κατά πολύ. Τώρα, για το ζήτημα της, της, της, τεχνολογίας πλάσματος. Αυτή είναι καινούρια τεχνολογία. Ε, Αλλά Ε, δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα κακής διοίκησης ή λανθασμένου συστήματος λήψης αποφάσεων που επελέγει αυτή η τεχνολογία. Κάθε τεχνολογία μπορούμε να δούμε πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα αλλά αν ένα, για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι έχει γίνει μια πολύ ε, εις αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν πολλοί και διαφορετικοί ε, ενδιαφερόμενοι φορείς στη Βουλγαρία, τα κρατημέλη ε, έδωσαν την άποψή τους, η Επιτροπή έδωσε την άποψή της, επομένως θα έλεγα ότι δεν ήταν αποτέλεσμα αυτή η επιλογή μιας χαόδους δομής λήψης αποφάσεων χωρίς λογοδοσία ή συντονισμό, δεν φταίει κάτι τέτοιο. Τώρα υπάρχουν ορισμένε αναφορέ ε, στην έκθεση που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν συμπεριληφθεί. Για παράδειγμα, αναφέρεστε στο Κοσλοντούι και λέτε. ότι εκατοντάδε ειδικοί εντό εισαγωγικών που ήρθαν από άλλα πυρηνικά εργοστάσια ανέλαβαν την, τον παροπλισμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζετε αυτά τα εισαγωγικά, δηλαδή τι σημαίνει ότι δεν ήταν ειδικοί. Πρόκειται για άτομα με εξαιρετικά υψηλά προσόντα και εξαιρετικά καταρτισμένα από τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, δεν καταλαβαίνω. Κάτι άλλο σημαντικό που αναφέρθηκε και προηγουμένω είναι το ζήτημα των καθυστερήσεων. Και πράγματι, ναι, υπάρχουν τέτοιε καθυστερήσει σε, διάφορες, σε διάφορα κράτη-μέλη, γιατί πρόκειται για μια νέα διαδικασία ε, και στα τρία από αυτά. Το ερώτημα όμω είναι, εάν υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρηση εξαιτία αυτών των καθυστερήσεων. Αυτό είναι σημαντικό για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε, να το εξετάσουμε περισσότερο, να λάβουμε υπόψη μα την εμπειρία του Κοσλοντούι, που είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο, του οποίου ο παροπλισμό καθυστερεί χωρί αυτό να επιφέρει επιπλέον κόστο. Και εξηγείται αυτό. Ωστόσο δεν καταγράφεται στην έκθεση ότι ο συνολικός χρόνος μέχρι, για τον παροπλισμό ενός πυρηνικού εργοστασίου μειώνεται. Δηλαδή έχουμε πάει από τα 20 στα 15 χρόνια και μειώνεται διαρκώς. Αυτό είναι γεγονός και ένα στοιχείο που δεν αναφέρεται στην εκθεσή σας. Με άλλα λόγια, έχουμε καταγράψει τα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν, ε, υπάρχουν διεστάμενες απόψεις από αυτόν, αλλά το ζήτημα που θα πρέπει εμάς να μα απασχολήσει είναι πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αν αυτό γίνεται με τον ορθό τρόπο. Αυτό πρέπει να συζητάμε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συναδέλφο Κάλβιν. Ναι. Θα ήθελα να πω πως εγώ τη συζήτηση αυτή θεωρώ πως δεν πρέπει να τη βλέπουμε ε, με την έννοια ότι έχουμε ένα ρόλο διαιτητή, λέει ο κύριος Γκάιερ. Ό,τι είναι από τη μία το Οικολογικό Ινστιτούτο και από την άλλη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανασυγκρότηση. Βεβαίω πρέπει να βγάλουμε τα πολιτικά μα συμπεράσματα, έτσι. Οπότε το τι τώρα έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα και το χρόνο, και τι ισχύει και δεν ισχύει, εντάξει, πρέπει να ξεκαθαριστεί. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα, το οποίο είναι σημαντικό για την πολιτική αξιολόγηση. Η ικανότητα της διοίκησης. Η Κομισιόν και η τράπεζα είπε πως ε, τα έργα αυτά είναι συγκρίσιμα γιατί οπωσδήποτε η διοίκηση στα τρία κράτη-μέλη τα οποία αναφέραμε δεν ε, είναι πολύ εξοικειωμένη και βεβαίως ε, θεωρούμε πόσο ε, ειδικά όσον αφορά τα κανένα κράτη-μέλη ε, υπάρχει μια κάποια δυναμία όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Α, εντάξει, κατανόηση όντως, αλλά δεν πρέπει όπως είπα να παραμελήσουμε και την πολιτική πτυχή. Οπότε εδώ πέρα το Οικολογικό Ινστιτούτο έχει μία αποστολή αλλά πρέπει να συγκρίνουμε και το τι συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη και το τι μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε για την κατάσταση αυτών των τριών κρατών μελών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή ανώμια πράγματα Δηλαδή η κάθε χώρα από αυτές τις τρεις έχει τη δικιά της ιστορία ε, βεβαίως ε, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με Γαλλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία που είχαν μια τελείως διαφορετική ιστορία με τα πολεμικά έτσι. Οπότε εντάξει ναι έτσι έχει η κατάσταση και πράγματι δεν είναι συγκρίσιμα, αλλά το ξέρουμε αυτό και θα ήταν και άδικο να πούμε πώς αναμένουμε στις χώρες αυτές να λειτουργούν τα πράγματα όπως σε Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία. Δεν γίνεται. Και αυτό βεβαίω θα μετρήσει στην πολιτική αξιολόγηση της κατάστασης. Εμάς λοιπόν είναι σημαντικό να πούμε με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και είδαμε και τις ε, καθυστερήσεις και την υπέρβαση του κόστους, ποιες δυνατότητες έχουμε να επιδράσουμε θετικά στην τράπεζα και στην ε, Κομισιόν, βεβαίω και στα κράτη-μέλη, να επιδράσουμε έτσι ώστε ε, να βελτιωθούν οι διαδικασίες επιτόπου για να αντιμετωπιστούν ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Και για εμάς ε, είναι σημαντικό και ένα άλλο θέμα. Αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν ως χρηματοδότηση. Στο επόμενο βήμα του παροπλισμού αρκεί ή μπορούμε από τώρα να βρούμε προβλήματα τα οποία θα καθυστερήσουν σαφώς ε, τα πράγματα και ε, θα κοστίσουν περισσότερο. Κατόπιν. Για την επιστημονική θεμελίωση της κουβέντας μας. Εδώ πέρα με τον κύριο Μαρινέσκο, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος εισηγητής, είχαμε έντονες διαφωνίες για το εάν η πολιτική θέση 2000, ε, για το 2020 πρέπει να συμβιβάζεται και αν είναι πραγματικά ρεαλιστική. Γιατί και για τη Σλοβακία που είναι αρκετά προχωρημένο το ένα έργο θα χρειαστεί τουλάχιστον μέχρι το 2028 να πάει. Και λένε κάποιοι συνάδελφοι, ναι εντάξει τότε θα σταματήσουμε τη χρηματοδότηση. Ε, ναι αλλά τότε δεν επιτυχάνουμε το στόχο έτσι της, ε, του παροπλισμού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία βάση και να πούμε το αναμενόμενο κόστος καλύπτεται. Στη Σλοβακία διαπιστώσαμε πως λείπουν 120 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται. Οπότε λέμε εντάξει να μπουν άλλα 120 εκατομμύρια στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην επόμενη επταετία μέχρι το 2020 αλλά εγώ θα ήθελα να δω εδώ πέρα τι τι ε, θα γίνει με αυτά τα 160 εκατομμύρια φτάνουν μετά υπάρχει και το θέμα που είπε η Ίγκε. Τι θα παραδώσουμε στο επόμενο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Ο κύριος Έρενχάουζερ. Α, έφυγε. Μάλιστα, ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας που πήγε στο Κοσλοντού, οπότε θα μιλήσω για αυτά που είδα. και την εντύπωση που αποκόμισα. Ε, κοιτάξτε, έχω... Μικτά, ανάμεικτα συναισθήματα. Η Βουλγαρία δεσμεύτηκε πριν μπει πως τουλάχιστον εν μέρη θα παροπλήσει το συγκεκριμένο αντιδραστήρα. Εξακολουθούν να εργάζονται από αυτού. Ε, οι μονάδε 1 έω 4 έχουν βγει εκτό, 5 έω 6 αναμένεται και μετά υπάρχει και η μονάδα 7 και η Βουλγαρία βεβαίω λαμβάνει σοβαρά κονδύλια Αφενό για τον παροπλισμό ε, και ε, για την πάυση λειτουργία και για τον ολοκληρωτικό παροπλισμό μετά. Μιλάμε λοιπόν για αρκετά λεφτά τα οποία θα καλύψουν και τις απώλειες από την λειτουργία και την παροχή ενέργειας σε ολόκληρη την ε, ε, Βουλγαρία και υποτίθεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για έβρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ε, κτλ. κτλ. Η εντύπωση που είχα από όλες τις συζητήσεις ήταν πως η απόφαση παροπλισμού του πυρηνικού εργοστασίου ήταν κάτι το οποίο όλοι θεωρούν λάθος. Έτσι. Και μας ξεκαθάρισαν πως το πυρνικό αυτό εργοστάσιο είναι σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής ε, αυτάρκειας της Βουλγαρίας και θα αφήσει πίσω του ένα τεράστιο κενό. Οι δε καθυστερήσεις λοιπόν ε, που προέκυψαν Πάντα βεβαίω ε, δικαιολογούνται με διάφορα επιχειρήματα κατανοητά, αλλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι γνωστά εκ των προτέρων. Ικανότητες, ε, δυνατότητες, το τι απαιτείται για τον παροπλισμό. Έπρεπε να τα γνωρίζουν αυτά. Αλλά πάρα πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, το είπαν και οι προλαλήσαντες. Και όταν το 2012 έγινε μια συζήτηση στην ε, Βουλγαρία μήπως τουλάχιστον δύο από τις μονάδες ε, έπρεπε να τις ξανανοίξουν ε, για να έχουν ρεύμα. Και η κυβέρνηση απλά είπε πως έχουμε απλά μια πολιτική απόφαση και συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό μου και αυτό ήταν το μόνο που είχε να πει. Μου δείχνει πως ε, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει έτσι και πολύ σοβαρή θέληση. Όσον αφορά τις ευθύνες. Όπως σας είπα, ε, τις εντυπώσεις μου μεταφέρω. Και συναντήσαμε βεβαίως πάρα πολλούς ε, οι οποίοι είχαν ο καθένας ένα κομμάτι ευθύνης αλλά ο κανένας δεν ήταν συνολικά υπεύθυνος. Και αυτό μου θύμισε στην ε, Ανατολική Γερμανία όπου μεγάλωσα τα... του σοσιαλιστικού καθεστώτος εκεί πέρα. Και το βιβλίο του κυρίου Μπαρό, ο οποίο μετά βεβαίως απελάθηκε από τη χώρα ενός κανομολόγου, ο οποίο περιέγραψε το καθεστώ ως οργανωμένη ανευθυνότητα. Αυτό μου θύμισε και πολλά ερωτήματα δεν απαντήθηκαν. Δηλαδή το 2012 είχαμε την αρχή, την Σέραφη, η οποία παραδείγματος χάρη είχε οργανόγραμμα 600 ατόμων αλλά επιτόπου στο εργοτάξιο είδαμε 30 τόσα άτομα και μας λένε θα και θα. Μετά, οι ράβδοι του αντιδραστήρα πήγαν στη Ρωσία γιατί δεν μπορούσαν να αποθηκευτούν. Και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν τώρα, προσωρινή αποθήκευση ή οριστικό μέτρο. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ βεβαίως. Και μπορώ να σας αναφέρω μια ολόκληρη σειρά παρομοίων καταστάσεων. Με τα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν υποτίθεται για έργα ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας ή για εναλλακτικές πηγές ε, ενέργειας ε, και εκεί πέρα δεν μάθαμε τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Όταν ρωτήσαμε μία μικιό αν είχαν άλλες πληροφορίες ε, και εκεί πέρα πάλι πολύ αρνητικές απαντήσεις. Οπότε για μένα παραμένει η εντύπωση πως συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στη Γερμανία. Δηλαδή όταν τα λεφτά έρχονται απ' έξω από κάποιον άλλον ε, ε, υπάρχει απλά η ελπίδα πως ε, θα πάνε καλά τα πράγματα και άμα δεν πάνε καλά θα πούμε τα γνωστά μας επιχειρήματα και μέχρι τότε ποιος ή ποιος πεθαίνει. Και μην ξεχνάμε είχαμε και την ε, Τρόιχαντ έτσι, που είχε αναλάβει τις ε, κρατικές εταιρείε Ανατολικής ε, Γερμανίας η οποία υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε για λίγα χρόνια και μετά από καμιά δεκαετία μας ανακοίνωσε δεν τα καταφέραμε να τις ε, καθαρίσουμε όλες ή να τις κλείσουμε ή να τις πουλήσουμε πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε άρα ως ε, εταιρεία διαχείρισης και τα λοιπά και τα λοιπά και συνεχίζουν βεβαίως. Γεγονός λοιπόν είναι πως έχουν πάει ένα σωρό λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου εκεί πέρα και πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον τι γίνεται. vielen Ευχαριστούμε κύριε Τσέλερ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Σμιτ, θέλετε να απαντήσετε. Ε, θέλετε Θέλω να να σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες και μομφές ε, που ακούστηκαν. Ε, επιφυλάσσομαι να απαντήσω γραπτός ε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα πιο σαφή. Ειδικά δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα εντυπώσει όταν κάποιο δεν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο με τι λεπτομέρειε και δεν έχει κανένα νόημα να μπω σε λεπτομέρειε. Τώρα ευχαρίστω όμω θα σα στείλω και να απαντήσω γραπτός χωρίς χρονικό όριο. Νομίζω πως προέκυψε και γι' αυτό είμαι ευγνώμων το ότι εμείς θέλαμε ακριβώς να προτείνουμε βελτιώσεις ε, ή να κάνουμε κάποιες προτάσεις βελτιώσεων. Βεβαίως δεν μπορούμε ε, εμείς να κάνουμε φτιάξουμε κανόνες έτσι για την κοινή χρηματοδότηση του παροπλισμού. Εάν θα θέλατε κάτι τέτοιο και αν το θεωρείτε αποτελεσματικό δηλαδή τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο τότε πραγματικά θα υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί ένα κίνητρο έτσι ώστε η χώρα η οποία ε, κερδίζει από αυτές τις επιδοτήσεις να φροντίσει και τα δικά της, να είναι και προς το συμφέρον της να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική. Αυτή είναι μία ε, ιδέα από αυτές που προτείναμε ακριβώς για να επιτύχουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο δηλαδή μόλις ο κύριος Τσέλερ περιέγριψε ως ε, οργανωμένη ανευθυνότητα. Πράγματι το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις στη Βουλγαρία αλλά και στην ε, Σλοβακία είδαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Και πραγματικά η οργάνωση νομίζω θεωρεί, ο οργανισμός εκεί πέρα θεωρεί πως ε, ε, αυτή είναι η βασική της αποστολή, ο παροπλισμός. Τώρα, το εάν αντιμετωπίζει τα ζήματα με κάποια αφέλεια ή κάνει αξιόπιστη διαχείριση κινδύνου και προβλέπει και κιόλας και προγραμματίζει, ε, εντάξει, ομολογουμένως εκεί πέρα υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Γιατί δεν πρέπει κανείς βέβαια να είναι αφελής και μετά να διαπιστώνει με έκπληξη ότι τα πράγματα πήγαν αλλιώς. Αν κάποιος έχει ως ε, φιλοσοφία εταιρική ή ως ε, επιχειρηματική αρχή κάποια πράγματα, συνήθως εκπλήσεται δυσκολότερα. Ή δεν έχει τόσες ε, καθυστερήσεις. Οι προτάσεις που κάνουμε λοιπόν είναι πράγματα που τα έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Τώρα, το εάν τα αντιγράψαμε από εγχειρίδιο οικονομικών, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ μου εγχειρίδιο οικονομικών, έτσι. Απλά βασίστηκα στο να κάνω κάποιες λογικές ε, προτάσεις, τίποτα παραπάνω. Αν είναι τώρα από εγχειρίδιο, τι να σας πω, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Είναι πράγματα τα οποία έχουν προκύψει από την δική μας την άμεση συμμετοχή σε ε, περιπτώσεις παροπλισμού και από τις συζητήσεις. Και βεβαίω υπάρχουν ε, πράγματι επιφυλάξεις που αναφέρατε για το εάν τα λεφτά αυτά είναι προς το συμφέρον του ε, Ευρωπαίου φορολογούμενου και αν χρησιμοποιούνται σωστά. Ε, σε αυτό σκοπεύει να συνεισφέρει η πρότασή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να βρίσκεται εδώ πέρα και ο εκπρόσωπος... Α, είναι εδώ πέρα. Ο εκπρόσωπος της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο κύριε Πίτορα. Θα ήθελα να κάνω, να μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο για τις αναλύσεις τις οποίες ακούσαμε. Οι Σλοβακικές αρχές προχωρούν στους ελέγχους που περιγράφονται και στην έκθεση είναι περίπλοκο το θέμα, δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να σας δώσουμε πλήρη σχόλια, αλλά θα σας στείλουμε τα σχόλιά μας σαν γραπτά τις επόμενες μέρες. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τώρα εάν το ελεκτικό συνέδριο θέλει να πει κάτι, όχι. Η Κομισιόν. Θέλει το λόγο ή είναι τα πράγματα σαφή. σε επίπεδο γενικό είμαστε στη διάθεσή σας για συζητήσεις ε, ή για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες. Επαναλαμβάνω ότι οι συστάσεις της εκθέσεως βασίζονται σε πάρα πολλές αμφισβητούμενες υποθέσεις. Αυτό έχει σημασία για μας. Κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε για τα αποτελέσματα της έκθεσης. Αλλά είμαστε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες και γραπτές επίσης, γραπτά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεσή σας και ενδιαφερόμαστε και για τις περαιτέρω εργασίες. Κύριε Ισηγητά, ναι, για να συνοψίσω, δεν έχει τελειώσει εδώ πέρα η υπόθεση. Επισκεφθήκαμε τις τοποθεσίες. Είδαμε τη μελέτη του Οικολογικού Ινστιτούτου. Οπωσδήποτε θα δούμε και με τις εθνικές αρχές σε ποιο βαθμό υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν οι συστάσεις του Οικολογικού Ινστιτούτου και βέβαια να βγάλουμε και τα πολιτικά μας ε, συμπεράσματα. Να δούμε ποια είναι τα ανοιχτά ακόμα ζητήματα και οπωσδήποτε πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ολοκληρωθεί η δουλειά μας εδώ πέρα, αν θα είναι μια έκθεση πρωτοβουλία στο επόμενο έτος Γιατί όποτε φαίνεται ε, η έκθεση πρωτοβουλία ανέδειξε περισσότερα ερωτήματα από αυτά τα οποία απάντησε, αλλά βεβαίω ε, υπάρχουν δύο αρμόδιες επιτροπές, η Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην οποία είμαστε πολλοί από εμά. Και βεβαίως ε, αυτό μας έδωσε την δυνατότητα ε, να δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί η εκταμίευση των 816 ε, εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια να βγάλουμε τα σχετικά μας συμπεράσματα και η Επιτροπή Βιομηχανίας βεβαίω. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Η απαλλαγή της Κομισιόν επίσης ε, μας δίνει μια ευκαιρία, αλλά δεν επαρκεί. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Τελείωσε αυτό το θέμα σήμερα στη μερίσια διάταξη. Το θέμα λοιπόν είναι ποια πολιτικά συμπεράσματα. Δεν να Ευχαριστώ για την Κομισιόν και για τη ειλικρινή τη ε, τοποθέτηση και ευχαριστώ την κυρία Στοχάλοβα και τον κύριο Σμιτ. Λοιπόν, τα ξαναλέμε στι 3. Γεια σας.